Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε καθυστερήσει και εγώ άργησα να φτάσω. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τις 5 και 4 έχουμε διερμηνία. Γιατί η διερμηνία χρειάζονται για τη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή, που βέβαια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δύο ώρες λιγότερες από ό,τι προβλέπεται κανονικά. Η κυρία Αλφάνο, που δεν είναι εδώ, όμως έχει ζητήσει να προσθεθεί ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη για την τακτοποίηση των μεταναστών στην Ιταλία. Προτείνω την επόμενη φορά να το δούμε, στην επόμενη συνεδρίασή μας. Οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα, εκτός αν έχετε παρατηρήσεις. Κλοντ. Η κυρία Αλφάνο θέλει να συζητηθεί στους συντονιστές την επόμενη συνεδρία των συντονιστών τη Δευτέρα, έτσι. Εκεί να το δούμε. Εντάξει, εντάξει, λέει η κυρία Σοφία Χιτφέλτ. Δεν βλέπω εδώ όμως κανένα συντονιστή άλλον εκτός από τον εαυτό μου. Όταν κανένας δεν είναι εδώ, τι γρήγορα που πάνε τα πράγματα και απλά. Φτάνουμε στο σημείο 3. Θέσπιση ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον ε, δικαστικό χωρισμό. Θα θυμόσαστε ίσως ότι δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη και περάσαμε στη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία. Την κυρία Κέπαρτ που είναι. Άνατη. Οπότε, κύριε Κέπαρτ, θα σα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που θα συζητήσουμε σήμερα το θέμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, γιατί πρόκειται για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που θέλουν να χωρίσουν και πολλές φορές έχουν τεράστιες δυσκολίες ε, να βρουν ε, το δίκιο τους στην ε, περίπτωση αυτή. Επειδή λοιπόν υπάρχει, υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά συστήματα στην Ευρώπη και η κατάσταση αλλάζει. Ε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να χωρίσουν αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είχαμε προσπαθήσει προετών να αλλάξουμε μία οδηγία όπου προστατεύονται αυτά τα δικαιώματα αλλά δεν ήταν δυνατόν να επιτύχουμε στο Συμβούλιο ομοφωνία και ξέρετε ότι ε, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ακόμη και με τη ε, συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των Υπουργών Δικαιοσύνης και δεν ήταν δυνατόν. Τώρα λοιπόν τον ε, Ιούνιο το, πολιτικό, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι μπορεί να υπάρχει και στην Ευρώπη μία διαδικασία μεταξύ κρατών μελών. Μία διαδικασία η οποία θα είναι μάλλον διακυβερνητική. Αλλά εν περιπτώσει εγώ είχα ζητήσει από την επιταγή, από την ε, ε, Επιτροπή και ε, το είχαμε συζητήσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα δεχόμαστε μία τέτοια διαδικασία διότι δεν έπρεπε να τεθεί ένα θεσμικό θέμα για κάτι το ουσιαστικό και το Συμβούλιο ε, μας είχε διαβεβαιώσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συζητήσει θα εμπλέκεται, πράγμα το οποίο θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητο. Εφόσον λοιπόν έθεσε το ερώτημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, συνένεσε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, βλήθη ε, από την Επιτροπή ένα κείμενο το οποίο ήταν θετικά εκπληκτικό δηλαδή για πρώτη φορά στην πρώτη διαδικασία το 2007-2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να αντικατοπτρίζεται στην απόφαση και την πρόταση που θα διατύπωνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίω όσον αφορά τα πιο δύναμα άτομα σε μία σχέση. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υιοθέτησε και αν το αξιολογώ σωστά είναι και ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί θετικά στο Συμβούλιο, δηλαδή είναι κάτι το θετικό που μπορούμε να πούμε ότι ναι, η προεργασία την οποία κάναμε αναγνωρίζεται και το αντικατοπτρίζεται ιδίως στα εκτιμώντας 13, 14, 15 όπου ε, λέγεται ότι οι δικαστές ή οι αρχές που πρέπει να αποφασίσουν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι και οι δύο εταίροι θα πρέπει να συμφωνήσουν για το δίκαιο ε, ε, υπό το οποίο θα γίνει, η διαδικασία. Και γι' αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη μεγάλες τροπολογίες. Οι τροπολογίες τις οποίες έχω περιλάβει είναι γενικώς διευκρινήσεις. Ιδίως όσον αφορά παραδείγματο χάρη τη σειρά στην ε, επιλογή ε, των ε, δικαίων βάση των οποίων θα ληφθεί η απόφαση δηλαδή ε, αν θα πρέπει να είναι η έννοια της συνήθους διανομής και ό,τι σημαίνει ή η μη διάκριση πρέπει να παίζει μια, ένα ουσιαστικό ρόλο σε αυτό το οποίο θα πράξουμε. Συνολικά λοιπόν έχω ίσα ίσα 8 τροπολογίες τις οποίες έχω καταρτήσει αλλά έχουμε ένα σύντομο πρόβλημα. Δηλαδή, το Συμβούλιο ε, θέλει τώρα να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να, ε, να εργαστούμε και στην Επιτροπή μας ε, πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σκιώδη Συγητή ε, και τους υπόλοιπους Σκιώδης Συγητές που προσαρμόστηκαν διότι εγώ διατύπωσα τις τροπολογίες μου αγγλικά ώστε στη συνάντηση των Σκιωδών Συντονιστών να μπορούμε να συζητήσουμε και η τροπολογία για τις, οι προθεσμοί για τις τροπολογίες είναι για μεθαύριο για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 29 Δεκεμβρίου διότι η Επιτροπή ε, της, ε, των νομικών υποθέσεων θα ε, ψηφίσει στις 2 Δεκεμβρίου και πρέπει να κινηθούμε πολύ ταχεία και ε, εφόσον λοιπόν δεν χρειαζόταν τόσο προεργασία όπως άλλα θέματα που κοίταξε η Επιτροπή, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη οθετήσει πολλά από αυτά τα οποία είχαμε διατυπώσει. Σκέφτομαι και θα ήθελα, πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την εξαιρετική εργασία την οποία έκανε. Γι' αυτό και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο έχουν να πούν επί του θέματος οι άλλοι σκιώδεις εισηγητές, εν που βρίσκονται εδώ σήμερα βέβαια. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να παρέμβει. η κυρία Αντζελίλη. Προηγουμένως όμως, κοιτάξτε πριν πάρετε το λόγο, δεν το είπα και σε εσά, αλλά σε όλους το λέω τώρα. Παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δίκαιο τα τελευταία θέματα στην εμερήση διάταξη να τα εξετάσουμε μόνο με τα αγγλικά. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να έχουμε τελειώσει πριν τις 5.30. Κύριε Αντζελίλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα είμαι σύντομη. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο που επετέλεσε και συμφωνώ στην θετική της αξιολόγηση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερα ισχύει αυτό φυσικά για την διασφάλιση των δικαιωμάτων ε, του πιο αδύναμου μέρους και πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία των, των πιο αδύναμων. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι εμείς θα έπρεπε ίσως με κάπως μεγαλύτερη σαφήνεια να ε, διατυπώσουμε και να πούμε τι θα γίνει τώρα με τους ανήλικους. Τι θα συμβεί με τους ανήλικους. Αν υπάρχει μια αντιπαράθεση, μια σύγκρουση των δύο γονέων σαν συνέπεια μιας, ενός διαζυγίου ή ενός χωρισμού, τότε ιδιαίτερα πλήττονται τα παιδιά φυσικά. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ακριβώς αυτό το, στην χάτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των ανήλικων σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση για άλλη μια φορά να αναφέρεται η δυνατότητα να υπάρχει μια διαμεσολάβηση στην οποία θα κατέφευγαν, ώστε ενδεχόμενα κάποιες διαφορές απόψεων ειρηνικά να μπορέσουν να επιληθούν πριν από το διαζύγιο φυσικά. Και αυτή η διαμεσολάβηση να μπορεί να οδηγήσει στο να αρθούν τέτοιου είδους συγκρούσεις. Και η 52 του 2008, αυτή η οδηγία δηλαδή, ρυθμίζει το αστικό πεδίο, το αστικό πλαίσιο και το οικονομικό πλαίσιο για αυτή τη διαμεσολάβηση και την δυνατότητα της διαμεσολάβησης στο οικογενειακό αυτό πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω αυτή η πτυχή ίσως πιο έντονα να εκπονηθεί, να διατυπωθεί από μας, να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα. Ίσως μπορεί η συγγήτρια να το λάβει αυτός πρόταση υπόψη και να θα υπάρξει και μια τροπολογία που θα κατατεθεί σχετικά. Κύριος Χέμαντς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα θέλατε να παρέμβετε. Α, η κυρία Κέλλερ όμως πρώτα, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και φυσικά πρέπει να πω ότι έχω μία ερώτηση. Απλά κάτι το οποίο δεν κατανοώ απόλυτα και ίσως μπορεί να επεξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί απέκλεισαν την ε, ε, γιατί ε, η αναφορά της ακύρωσης ε, του γάμου και αν κατανοούμε ότι θα υπάρξει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011, όμως αυτό συνδέεται πολύ στενά με το ζήτημα αυτό και θα ήταν πάρα πολύ κρίσιμο, κέρια σημασία να ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση θα πορευθεί αυτή η πρόταση για να γνωρίζουμε κατά το μάλλον τον τι θα αναμένουμε. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν. Όχι, κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, πολύ καλά. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα μου. Και απλά μπορώ να επαρκεστώ και να πω ότι υιοθετώ τη δική σας γραμμή. Δεν νομίζω ότι θα κατατεθούν κάποιες τροπολογίες. Ίσως μία ή δύο όλες όλες. Αλλά θα ενισχύσουν τη δική σας αυτή, ας το πω έτσι, θέση. Τώρα η συγγύτρια και πάλι αν έχει κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις να κάνει. Η κυρία Γκέπαρτ, ευχαριστώ. Το θέμα της μέρημνάς σας στην οδηγία στο 3α ή όπως και να το αποκαλέσουμε αυτό το εδάφιο ρυθμίζεται εκεί και γι' αυτό δεν έχει κάποια άμεση σχέση με αυτό, αλλά όμως αν σε μια αιτιολογική σκέψη, σε ένα considerant μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτή η πρόταση ώστε να αποσαφινιστεί αυτό, κύριε, από πλευρά Αντζελίλη συμφωνώ απόλυτα να υπάρξει μια τέτοια αναφορά. Να καταθέσετε μια τέτοια τροπολογία παρακαλώ δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην, γιατί να μην υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Όταν πρόκειται για διαζύγιο, οι πιο αδύναμοι, ιδιαίτερα τα παιδιά πρέπει να προσέξουμε τι θα απογίνουν. Και αυτό ήταν εκείνο και το οποίο εννοούσα τότε στο παρελθόν όταν είχαμε την έννοια της προστασίας των πιο αδύναμων στο γάμο. Όχι των πιο αδύναμων απλά και μόνο στον γάμο αλλά και να δούμε τι συμβαίνει με την περίπτωση της ε, μέρημνας ε, παιδιών και το τι μπορεί να γίνει. Και καλό είναι μια τέτοια επισήμανση να μπορεί να ε, ενταχθεί εδώ. Ω αιτιολογική σκέψη όμως. Δεν νομίζω ότι στα άρθρα μπορεί να ενταχθεί αυτό. Διότι είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα από αυτό το οποίο έχουμε να διαβουλευτούμε εδώ. Αλλά καταρχήν να ληφθεί υπόψη αυτή η ιδέα θα το χαιρέτιζα και μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Και το θέμα της κυρίας Κέλλερ Λυπούμε, δεν το κατάλαβα πολύ καλά τι θέλατε να μάθετε, γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Ευχαριστώ. You want to raise your question again, or... Θέλετε να ξαναδιατυπώσετε το ερώτημα, κυρία Κέλλερ, ή μπορεί διμερώς αυτό να αποσαφινιστεί. Η ερώτηση ήταν γιατί ακύρωση γάμου. Γιατί δεν εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτή η έννοια. Εντάξει, διμερώς θα το συζητήσετε και θα αποσαφινιστεί αυτό. Περνάμε στο 4 στην ημερήσια διάταξη. Θα ζητήσω από όλους τους εισηγητές και τα μέλη που να λάβουν το λόγο για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα θέματα. Οι εισηγητές σε τρία λεπτά θα πρέπει να παραμείνουν στην παρέμβασή τους, στην αρχική τους παρέμβαση και τα μέλη της Επιτροπής μας θα παρεμβαίνουν για ένα λεπτό και να δούμε πόσο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Επόμενο θέμα η ενίσχυση όσον αφορά τα θέματα χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκίτρια και Γκόμες θα έπρεπε να πω προηγούμενα να αναφέρω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι μεθαύριο και θα ψηφίσουμε στις 29. κυρία Γκόμες έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η έκθεση που έχετε μπροστά σας στα χέρια σας έτυχε 123 τροπολογιών. Και εγώ η ίδια ως εισηγήτρια κατέθεσα 41 από αυτές τις 123 τροπολογίες. Και αυτές οι 41 τροπολογίες απέρευσαν από τις προσωπικές μου επαφές με επαΐοντες, πραγματογνώμονες, οργανώσεις και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμούς και υπηρεσίες και όσον αφορά και θέματα που αφορούν και την Πορτογαλία, τη χώρα μου, μια και είναι γνωστό ότι δεν είναι μια από τις χώρες όπου οι διεργασίες και οι διαδικασίες να είναι οι πιο αυστηρές για αυτά τα θέματα για την ραδιολογική, χημική, βιολογική προστασία και την προετοιμασία κατά των ε, επιθέσεων όσον αφορά τις βιολογικές πτυχές, ραδιολογικές, χημικές, πυρηνικές, αλλά δεν είναι και η χειρότερη χώρα όσον αφορά την προετοιμασία της για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων και εξεπλάγει βλέποντας ότι έχοντας ακούσει όλες τις, όλους τους οργανισμούς σε δημόσια κρόση εξεπλάγει ότι βρήκα και τελικά διαπιστώθηκε ότι όλοι ήξεραν για το πρόγραμμα δράσης όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα δράσης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο πριν από ένα χρόνο και υποτίθεται ότι από τον προηγούμενο Ιούλιο υλοποιείται και όλοι οι οργανισμοί στην χώρα μου, την Πορτογαλία, είχαν συνειδητοποιήσει και γνώριζαν αυτό το πρόγραμμα δράσης και κάποιοι οργανισμοί συμμετείχαν ε, δραστήρια και στη διατύπωση όλων αυτών, αλλά ταυτόχρονα δεν υλοποιούνται, δεν υλοποιούνται όλα αυτά. Και αυτό είναι το χειρότερο σε σχέση με το αν δει κανείς τι γίνεται στα κράτη-μέλη με το πώς αντιδρούν για αυτά τα θέματα. Φυσικά γνωρίζοντας ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες και είναι αποτέλεσμα είτε φυσικών καταστροφών είτε σαν εκείνη την τοξική μόλυνση των ποταμών στην Ουγγαρία με την τοξική λάσπη ή τρομοκρατικές επιθέσεις όπως είδαμε και πρόσφατα με αυτά τα πακέτα, τα δέματα που είχαν αποσταλεί από το ταχυδρομείο με ε, κάποια, κάποιες ε, χημικές ουσίες, σκόνες κτλ δεν είναι πραγματικά πρέπει να πούμε καταστάσεις ε, απλά χαμηλού κινδύνου και πρέπει να προετοιμαστούν οι χώρες μας και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κέρια σημασίας και η δημοσίευση αυτής της έκθεσης στοχεύει στο να ενισχυθεί αυτή η πτυχή της προστασίας και να ενισχυθεί η ρυθμιστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει τα κράτη-μέλη. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε το δυναμικό των κρατών μελών κέριο, κύριο συμπέρασμα, δεν θα επισέλθω σε όλα, αλλά ένα κύριο συμπέρασμα που αποκόμισα από την ακρόαση που κάναμε στην Πορτογαλία, τη χώρα μου, είναι ότι οπωσδήποτε χρειαζόμαστε σε εθνικό επίπεδο μια υπεύθυνη αρχή για την διατύπωση και συντονισμό όλων αυτών των συστάσεων και την επιτήρηση των άλλων ε, υπηρεσιών που εμπλέκονται από το, τη δημόσια υγεία για την πολιτική προστασία κτλ. Διάφοροι εμπλέκονται, αλλά αν δεν συντονίζονται από κάποιον και δεν διαχέονται οι πληροφορίες, τότε δεν θα είναι αποτελεσματική προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Ε, υπήρξαν τροπολογίες που καταρτίστηκαν και ουσιαστικά μπορώ τις περισσότερες από αυτές να δεχθώ, διότι πραγματικά προσθέτουν αξία και περιεχόμενο στην έκθεση δεν βρίσκονται με κανένα τρόπο σε αντίφαση με αυτά τα οποία πρότεινα και ήθελα να, να προτείνω εγώ. Δύο σημεία όλα και όλα, όχι σύγκρουση συμφερόντων ή κάποιας ε, ε, διαφοράς, αλλά σε μια συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές είδαμε ότι υπάρχουν δύο ευαίσθητα κύρια θέματα. Έχω ε, προτείνει διατυπώσεις ε, συμβιβαστικές και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν δεκτές. Δεν θα είναι δύσκολο φαντάζομαι αυτό το σημείο. Βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματος. Πιθανότατα το ε, μόνο διακόπτη πρόεδρος θα ήθελα να ολοκληρώσετε. Γι' αυτό πρότεινα συμβιβαστικές τροπολογίες για να δούμε αν η βιομηχανία ή όχι θα μπορούσε να αναλάβει την πληρωμή, την κάλυψη του κόστους της υποκατάστασης ή επικίνδυνων ουσιών, δηλαδή κυρίως χημικών ουσιών ή άλλων τέτοιων ουσιών, όταν αυτό τεχνικά μπορεί να γίνει και επιστημονικά είναι εφικτό. Έχω διατυπώσει με τέτοιο τρόπο αυτές τις προτάσεις που δεν είναι τόσο ριζοσπαστικές όσο οι αρχικές μου προτάσεις και οι συνάδελφοι που είχαν πρόβλημα με αυτές τις ριζοσπαστικές ε, προτάσεις μου τώρα δεν θα έχουν πια. Θα ψηφίσουμε στις 25 Νοεμβρίου στην έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Δύο ζήτησαν τον λόγο ο κύριος Άλβαρο ο κύριος Πανός και κάποιοι άλλοι. Ο κύριος Άλβαρο, παρακαλώ. Όλοι ένα λεπτό παρακαλώ, συνάδελφοι, να είσαστε σύντομοι και περιεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Άννα. Μιλάω εκ μέρου τη Σεσίλια Βίλστρομ ουσιαστικά, που είναι σκιώδη εισηγήτρια για αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώ καθυστέρησε η πτήση τη και δεν θα μπορέσει να φτάσει έγκαιρα. Για αυτό το θέμα λοιπόν θέλω να αναφερθώ στις τροπολογίες της Σεσίλια που έχουν συζητήσει σίγουρα μεταξύ τους Άννα και Σεσίλια για μέτρα που να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τη σημερινή απειλή τρομοκρατία και με τις τροπολογίες αυτές θέλει και το κόστος να μειωθεί αλλά και η απειλή να μειωθεί και η αντίδραση να είναι αναλογική κάθε φορά. Η Σεσίλια στηρίζει τροπολογίες που μιλούν για έναν πιο σημαντικό ρόλο της Επιτροπής προκειμένου να φροντίσουμε για την ασφάλειά μας στο μέλλον. Σίγουρα έχει μιλήσει με την Ανακόμες και ότι άλλες συμβαστικέ τροπολογίες προκύψουν θα τις συζητήσουν μεταξύ τους οι δύο. Πρόεδρος, ωραία, ευχαριστούμε. Πέντε έχουν ζητήσει τώρα το λόγο. Ο κύριος Μπρόντς είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ. Ίσως ενδυνάμει να υπάρχει ένα πρόβλημα ε, από την χρήση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών, υπερηνικών παραγόντων από τους τρομοκράτες. Σήμερα πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι υπάρχουν δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεράσουν οι τρομοκράτες πριν να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τελικά αυτά. Η Επιτροπή πάντως και άλλοι δεν χάνουν ευκαιρία να επεκτείνουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας νέα σώματα, επεκτείνοντας τα υπάρχοντα σώματα και αναθέτοντας τους νέες αρμοδιότητες. Η, η συγγήτρια έχει καταφέρει να μειώσει το δεσμευτικό χαρακτήρα της σύστασης και μιλάει και για περιπτώσεις στρατιωτικής χρήσης. Η Επιτροπή δέχεται ότι δεν είναι εύκολο να οργανωθεί η αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής, όμως παρόλα αυτά λέμε ότι πρόκειται για σοβαρή ε, απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, συνενούνται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και μυστικές πληροφορίες αντί να δημιουργήσουμε ένα νέο σώμα, ένα νέο όργανο που θα είναι αρμόδιο για αυτή τη δουλειά. Ευχαριστούμε, κύριος Μπουσάτηλ. Εγώ θέλω να μιλήσω εκ μέρου τη κυρία ε, που είναι η σκιώδη εισηγήτριά μα. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ε, εισηγήτρια και να ξέρει ότι στηρίζουμε ευρέω την προσέγγιση τη. Και εμεί πιστεύουμε ότι η απειλή από τέτοιου ε, κινδύνου είναι όντω πραγματική. Συμφωνούμε λοιπόν με τον τρόπο που βλέπει το θέμα. Είναι αρκετά πλήρης η έκθεσή της. Λίγα πράγματα θα είχα να προσθέσω ή να διευκρινίσω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πρόθεση της ε, εισηγήτριας να υποβάλει συμβιβαστικές τροπολογίες με τις οποίες θα καλύπτονται όλες οι ανησυχίες όλων των πλευρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο Υπουργό Δεκλέρκ, εξ μέρου τη Ολλανδική Προεδρία, ήρθε, οπότε να τελειώσουμε με τους ομιλητές Δίας Δεμέρα και Μέλντερ, πολύ γρήγορα όμως παρακαλώ, για να περάσουμε μετά στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσία του εδώ. Λοιπόν, το πρόγραμμα δράσης για τους χημικούς, βιολογικούς, ραδιολογικούς και πυρηνικούς κίνδυνους έχει δύο πλευρές. Το ένα είναι εναντίον πιανού και το δεύτερο είναι για ποιο λόγο. Θέλουμε να αποφύγουμε φυσικές καταστροφές, θεομηνίες. Γιατί? Για να είμαστε έτοιμοι με την πρόληψη και με την αντιμετώπιση. Να είμαστε σε θέση να οργανώσουμε την αντίδρασή μας, αν έχουμε τέτοια απειλή. Άννα, 8 τροπολογίες έχω. Σε ευχαριστώ για τη δουλειά σου. Είναι δουλειά πολύ σημαντική που έχει κάνει και 8 τροπολογίες μου στόχο έχουν την συνεργασία μας για τη βελτίωση της έκθεσης αυτής. Θέλω όμως να χρησιμοποιήσουμε και έναν πιο σωστό ορισμό όταν μιλάμε για τους τύπους δραστηριότητας που μπορούν να θεωρηθούν σαν τρομοκρατικές ή που προωθούν τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη των κινδύνων όσον αφορά την χρήση των προϊόντων. Μιλάμε για χημικούς και άλλους που αναφέρονται στο ρίτς. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο και εντάξει 20 δευτερόλεπτα δώστε μου ακόμα. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε τις αρμοδιότητες συντονισμού για την προστασία των πολιτών που τις έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος Διακόπτη, ολοκληρώστε παρακαλώ. Η ευθύνη πρέπει να είναι μοιρασμένη και στα κράτη-μέλη, λέει ο μιλητής. Ευχαριστούμε. Κύριε Μίλντερ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καρδιά του ζητήματος ε, είναι το βασικό είναι ο συντονιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει ορισμένες ε, υποχρεώσεις και ευθύνες και πρέπει να τονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη περισσότερο το θέμα αυτή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να εξασκήσει τον έλεγχό του το Κοινοβούλιο όπως πρέπει. Ε, ευχαριστώ. Η συγγήτρια, ένα λεπτό. Θα ήθελα να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις των συναδέλφων ότι δεν προτείνουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σώμα. Θέλουμε να εξουσιοδοτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο, κάτι που είναι απολύτω απαραίτητο. Χρειάζεται συντονισμός και μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών αρχών διότι ε, ε, υπάρχουν περισσότερες ε, γνώσεις σχετικά με τις επιθέσεις οι οποίες να είναι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές. Και γι' αυτό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να επαφίονται στα θέματα αυτά εις ε, την ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα φύγω, αλλά θέλω να σας πω ότι στηρίζω πλήρως την επιστολή που έστειλε η Διεθνής Αμνηστία στον πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με την λογοδοσία, σχετικά με τις παραδόσεις υπόπτων στις Αμερικανικές αρχές. Το επόμενο θέμα ε, είναι η σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία ε, που είναι επανάληψη της απόφασης ε, πλαίσιο 2004, μάλλον αναθεώρησή της και κατάργησή της και δίνω το λόγο στην κυρία Εντζελίλη που είναι η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ φυσικά την Βελγική Προεδρία, ιδιαίτερα τον Υπουργό Ντεκλέρκ, ο οποίος ήταν ευγενικό και θα είναι στη διάθεσή μας το απόγευμα. Και βλέποντας και εξετάζοντας τη δουλειά από πλευρά του Συμβουλίου για την Οδηγία για την Αποφυγή Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων και σε σχέση και με την απόφαση του 2004. Ξέρω ότι το θεωρεί προτεραιότητα το Συμβούλιο αυτό το θέμα και γνωρίζω προφανώς ότι εξακολουθούν και υφίστανται κάποια κέρια κρίσιμη σημασία σημεία, κυρίως όσον αφορά τις διαφορές στα νομικά συστήματα, τα υφιστάμενα νομικά συστήματα και τις διατάξεις και κανονισμούς στα 27 κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζεται η δουλειά γίνεται δουλειά για να επιτευχθούν λύσεις. Εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διαδραματίσουμε το ρόλο μας και είμαστε πεισμένοι ότι με την επικοδομητική συνεισφορά όλων θα είναι εφικτό να επιτευχθεί μια θετική και ελπίζω ένα θετικό και μάλιστα κιόλα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο Στρασβούργο. Είχε παρουσιαστεί ένα έγγραφο εργασία και το οποίο θα ξεκινήσουμε να συζητάμε, θα υποβληθεί ένα έγγραφο εργασία και θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Νόημα όλο, όλο αυτού του εγχειρήματο είναι να παρουσιαστεί η έκθεση τον Ιανουάριο και να έχουμε αυτές τις πτυχές που θα αποσαφινιστούν και θα διευθετηθούν το Φεβρουάριο. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τη Βελική Προεδρία και να ευχαριστήσω για τη διαθεσιμότητα και παρουσία του Υπουργού σήμερα και θα ακούσουμε τις λεπτομέρειες από τον ίδιο τον Υπουργό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεκλέρκ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας σήμερα. Και νομίζω ότι όλοι εδώ είμαστε επιπισμένοι ότι πρόκειται για ένα θέμα προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει και για την Βελγική Προεδρία. Προσπαθούμε πραγματικά όσο γίνεται πιο γρήγορα να καταλήξουμε σε συμφωνία στο Συμβούλιο. Εννοείται ότι μας ενδιαφέρει η επίπτωση που έχει στα παιδιά η σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση. Καταστρέφεται η ζωή τους, μένουν σημάδια σε ολόκληρη τη ζωή τους από τέτοιου είδου πρακτικές. Γι' αυτό και πρέπει με κάθε τρόπο και κάθε είδους τέτοια κακοποίηση να την αποφύγουμε και να την καταπολεμούμε. Υπάρχουν μέτρα καταστολής βέβαια που υιοθετούνται Ξεκινήσαμε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία και ευχαριστούμε για την πρότασή της, που αναφέρεται στις διάφορες μορφές κακοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τις καταπολεμήσουμε, κάνοντας πιο αυστηρές τις κυρώσεις. Βέβαια, έχουμε σιγά σιγά συλλέξει εμπειρία και μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε βάσει της εμπειρίας αυτής. Όσο προτεραιότητα, Στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου έχουμε αυτό το θέμα, αλλά και κατά το παρελθόν στο Συμβούλιο συζητήσαμε για αυτά, τον Οκτώβριο για παράδειγμα, και ο στόχος μπορεί να φαίνεται απλός, αλλά να ξέρετε ότι τεχνικά και νομικά, δικαστικά δηλαδή μιλώντας, δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε να συντονίσουμε τους μηχανισμούς που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Πάντως, στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση των ορισμών πρώτα απ' όλα και δεύτερον ε, για το επίπεδο των ε, ποινών. Γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ε, παραβιάσεις διαφορετικού τύπου, διαφορετικού βαθμού και πρέπει να προσπαθήσουμε, είναι μεγάλη φιλοδοξία βέβαια, το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε και με τα βάση του κεκτημένου που έχουμε από το 2003 και με το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2007 που έκανε την σύμβαση του Λαθαρότε, με όλα αυτά τα στοιχεία να δουλέψουμε για να καθορίσουμε τα νέα μέτρα. Το τελευταίο στοιχείο τώρα είναι το ότι υπάρχουν και νέα στοιχεία τεχνολογίας που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τις διαφορετικές δικαστικές παραδόσεις ή τις διαφορές που υπάρχουν στα ήθη και έθιμα των χωρών. Το Δεκέμβριο πάντως θέλουμε να καταλήξουμε σε κάτι ώστε οι Ούγγροι συνάδελφοι να μπορέσουν μαζί σας από την αρχή της επόμενης χρονιάς να δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα. Προσπαθούμε λοιπόν τις συζητήσεις μας να τις χωρίσουμε σε δύο τμήματα. Η Πρώτη συζήτηση θα είναι γίνει για τα άρθρα έως 13 και ήδη τον Οκτώβριο προχωρήσαμε σε αυτό το σημείο πολύ. Τώρα μας μένει κυρίως το δεύτερο τμήμα, το οποίο θα γίνει το Δεκέμβριο. Συνοψίζοντας, το πρώτο τμήμα. Τι είναι η συζήτηση του πρώτου τμήματος. Έχει τρία στοιχεία, όπου η Επιτροπή έκανε προτάσεις. Και το Συμβούλιο πρέπει να προσαρμόσει το Συμβούλιο όσον αφορά τις κυρώσεις θέλει να υπάρχουν ε, ε, ισχυρές κυρώσεις αλλά να υπάρχει και κάποια αναλογία με τα άλλα μέσα που έχουμε στο δικαστικό μας δίκαιο. Για ορισμένα παραπτώματα το Συμβούλιο κάνει μια διάκριση ανάλογα με την ε, ηλικία ε, κατά την οποία έγινε η κακοποίηση. Και ανάλογα με την ηλικία κάνει κάποιες διαφοροποίησεις. Αυτό ήταν το πρώτο τον Οκτώβριο που συζητήθηκε. Το δεύτερο ήταν ότι θέλει να προσαρμόσει επίσης το Συμβούλιο ε, τα μέσα που χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει την κακοποίηση αν γίνεται μεταξύ ατόμων ίδιας ηλικίας, μεταξύ φίβων δηλαδή. Και σε αυτό το επίπεδο, όταν πρόκειται μεταξύ παιδιών ίδιας ηλικίας, να δούμε και εκεί τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν από την δίωξη ε, παιδιών αυτής της ηλικίας για σεξουαλικές κακοποίησεις. συζητήθηκε πολύ το άρθρο 13 που λέει ότι οι ανήλικοι θεωρούνται θύματα και γι' αυτό μπορεί να μην τιμωρηθούν τελικά, επειδή θεωρούνται θύματα. Θέλουμε να το δούμε όμως αυτό και σε σχέση με άλλες διατάξεις των νόμων που έχουν να κάνουν με την πορνογραφία. Αυτά για τον Οκτώβριο. Τι, συζητήθηκε τώρα, θα συζητηθεί μάλλον τώρα το Δεκέμβριο, που θα είναι η δεύτερη σειρά άρθρων από το 2013 και μετά. Εδώ πέρα πρόκειται για την διαδικασία, για την πρόληψη. Θέλουμε συνολικά να δούμε το θέμα στη συνέχεια. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή σωστά αντιμετωπίζει το θέμα συνολικά Ελπίζουμε λοιπόν ότι και η πρόληψη θα συμπεριλαμβάνεται εδώ. Πάντως υπάρχουν τρία στοιχεία στη συζήτηση. Δεν υπάρχει ακόμα καθορισμένη θέση, συζήτηση γίνεται στο Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τρία σημεία που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά για την προετοιμασία μας. Το ένα είναι το άρθρο 10 που μιλάει για την απαγορεύση δραστηριοτήτων με παιδιά σε ανθρώπους που έχουν ήδη καταδικαστεί. Αν κάποιος δηλαδή έχει ήδη καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση, να μην μπορεί να αναλάβει επαγγελματική δραστηριότητα με παιδιά. Πρέπει να τεθεί αυτή η αρχή, πιστεύουμε. Αλλά βέβαια το ερώτημα είναι πώς θα το πετύχουμε αυτό. Τι μέσο θα έχουμε στη διάθεσή μας για να το πετύχουμε. Ε, γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάτι οριζόντιο. Πάντως γεγονός είναι ότι την αρχή αυτή την θέλουμε. Και την αναγνώριση των ε, καταδικών σε μια χώρα από άλλες χώρες για να μπορεί εύκολα να εντοπιστεί ένα τέτοιο άτομο και να μην μπορέσει σε μια άλλη χώρα να αναλάβει επαγγελματικά δραστηριότητες με παιδιά. Άρα λοιπόν θέλουμε αυτή την αρχή. Η συζήτηση εξακολουθεί να γίνεται, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε πώς θα έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίες οι αρχές δηλαδή που θέλουν να προσλάβουν τέτοια άτομα, πώς θα έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για να ξέρουν τι έχει γίνει στο παρελθόν. Ενημέρωση δηλαδή του εργοδότη. Αυτό είναι κάτι που πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδες. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα γίνει στη... που θα συμπεριληφθεί στη συζήτηση του Δεκεμβρίου. Δεύτερον, πώς μπορούμε αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε τον σεξουαλικό τουρισμό Το Συμβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη του και τα διαφορετικά δικαστικά συστήματα που υπάρχουν στις χώρες, τις διάφορες, γιατί στο Βέλιο μπορεί να γίνει αυτό, σε άλλες χώρες ίσως όχι. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε έναν αποτελεσματικό τρόπο ώστε τέτοιου είδους σεξουαλικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό να καταπολεμηθούν. Και το τρίτο, και δεν θα σας εκπλήξει, είναι πώς θα μπλοκάρουμε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο πορνογραφίας. Με ποιο τρόπο μπορούμε να εμποδίσουμε την εμφάνιση τέτοιων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Είναι ευαίσθητο θέμα αυτό, για το οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Εγκατακλείδη. Ελπίζουμε με αυτό το ρυθμό να προχωρήσουμε γρήγορα Είπαμε, υπάρχει το πρώτο τμήμα που εξετάστηκε τον Οκτώβριο, το δεύτερο τμήμα θα εξεταστεί το Δεκέμβριο. Σας είπα ποια είναι τα τρία κρίσιμα σημεία που θα συζητηθούν ε, δίχως άλλο. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και ελπίζω ότι θα έχουμε τριμερή διάλογο με το Κοινοβούλιο και με την ε, Κομισιόν που να οδηγήσει σε αποτελέσματα ικανοποιητικά για όλους. Είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια αυτή που κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό δικαστικό μέσο που θα έχουμε στην διάθεσή μας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε σας σήμερα. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την εισαγωγή παρουσίαση. Και τέσσερις έχουν ζητήσει τώρα τον λόγο στη συνέχεια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να είσαστε σύντομοι, αν γίνεται, διότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. Υπάρχει καθυστέρηση χρονική όσον αφορά το αρχικό χρονοδιάγραμμα και ακόμα πιέζει περισσότερο χρόνο σε σχέση με το νέο χρονοδιάγραμμα. Να είσαστε αλληλέγγυοι και σύντομοι. Αλβάρο πρώτα. Ευχαριστούμε την, ε, για την παρουσίαση και ευχαριστούμε την κυρία Αντζελίλη για το έργο της και για την παρέμβαση εξ ονόματο της κυρίας Βίξτρομ. Ξέρω ότι υπάρχουν μέλη που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και εγώ ενδιαφέρομαι. Σε σχέση με αυτά τα θέματα είχαμε συζήτηση πέρυσι για αυτά και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα θέμα το οποίο έχουμε εδώ ενώπιον μας και για τα άλλα επίμαχα θέματα που σίγουρα υφίστανται σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω αυτό ειδικά. Η Επιτροπή Πολιτισμού ψήφισε τη γνωμοδότησή της και ήταν ομόφωνα υπέρ της πρότασης να αναζητηθεί η διαγραφή των ιστοτόπων που διαχέουν τέτοιου είδους υλικό όσον αφορά την κακοποίηση παιδιών. Ευθυγραμμίζομαι με άλλους συναδέφους ότι η πορνογραφία για αυτού του είδου το υλικό είναι κάπως ε, μια παρανόηση ή κάπως παραπλανητική. Διότι εδώ πρόκειται για την κακοποίηση και την κακομεταχείριση των παιδιών με το χειρότερο τρόπο. Όμως σε σχέση με την κατάργηση αυτών των ιστοτόπων είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε βέβαια αν θα πρέπει να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι αποτελεσματικά στα μέτρα που θα υιοθετούν ώστε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή και αυτό το πρόβλημα το να υπάρχουν φραγές ε, στους ιστοτόπους δεν φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσματικό διότι εξακολουθεί να υφίσταται το θέμα της πορνογραφίας όσον αφορά τα παιδιά. Κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν ε, έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο πρόσφατα είπε και είναι ίσως ενδιαφέρον αυτό και αναφέρω παράθεμα ότι θα πρέπει να ζητηθεί από τις ΗΠΑ ή τη Ρωσία να, να διαγράψουν, να απαλείψουν κάποιους ιστοτόπους ε, από το διαδίκτυο. Αυτό όμως ε, δεν έχει κάποια πρακτική επίπτωση, διότι αυτές οι χώρες δεν είναι πρόθυμες να κάνουν κάτι τέτοιο και για διάφορους ε, λόγους κιόλα. Και θα ήθελα και πάλι να ζητήσω, να ρωτήσω από την Προεδρία Πόσα κράτη-μέλη θα ήταν υπέρ μια τέτοια προσέγγιση να αποφασίζουν τα ίδια τα κράτη-μέλη αν θα θέλουν να επιβάλλουν φραγέ ή να διαγράφουν, να απαλήφουν από, τον ιστο... από το διαδίκτυο τέτοιου ιστοτόπου. Πρόεδρο, παρακαλώ να είστε πιο πειθαρχημένοι συνάδελφοι. Αλλιώ οι άλλοι συνάδελφοι δεν θα έχουν χρόνο να παρέμβουν. Δεν φταίω εγώ για το ότι πιέζει τόσο πολύ ο χρόνο. Αν όλοι κάνετε μια προσπάθεια θα ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Κύριος Μπρόνς παρακαλώ μετά. Υπήρχε μια κρόαση στην αρχή Οκτωβρίου και ήταν τόσο ε, αραιή η συμμετοχή που δεν ε, ε, μπόρεσε να τύχει συνέχεια. Υπήρξε εκπρόσωπος της ΜΟΓΕΣ οργάνωσης συλλόγου θυμάτων και αυτή η οργάνωση ήταν κατά της τροχοπέδης, ας το πω, της φραγής σε τέτοιου είδους ε, ιστοτόπους. Είπαν ότι είναι απλώς ένα εξοραϊστικό μέτρο η επιβολή τέτοιων φραγών. Και πάλι ο όρος ε, παιδική πορνογραφία μπορεί να είναι παραπλανητικός ε, ή όταν πρόκειται για κακοποίηση παιδιών με τέτοιου είδους εικόνες. Πιο συνήθιστο ήταν ότι υπήρχε ένας εκπρόσωπος ε, όσον αφορά κιόλας και την Ιρλανδία τονίζοντας ε, μια πτυχή του προβλήματος που εγώ δεν γνώριζα ότι υπήρχε. Και αυτό είναι ότι δεσμεύουν, σε, ε, συνδέουν αυτού του είδους τους ιστοτόπους σε κάποιες νόμιμες δραστηριότητες επιχειρήσεών τους. Και αυτό γίνεται πολλές φορές χωρίς άλλοι να το γνωρίζουν και χωρίς ε, να το θέλει κανείς ξε, είναι έτσι ξενιστή ας το πω έτσι πάροχος ε, τέτοιου είδους ε, πληροφοριών και εικόνων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εγώ δεν θα επισέλθω στα θέματα ουσίας, αλλά κυρίως στην διαργασία, στη διαδικασία για την επιβολή φραγών ή εμποδίων. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο μια αντιπαράθεση με νομικές παραδόσεις εδώ, ή κάποια ευαίσθητα θέματα. Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση. Πολιτικό θέμα. Αν θέλει κανείς να επιβάλλει φραγές παράλληλα με την διαγραφή και εξάλληψη ή απάλληψη ή όχι. Και ακούω επανειλημμένα ότι δεν λειτουργεί λέει αυτή η απάλληψη ή διαγραφή. Διότι σε σχέση με συνεργασία με τα κράτη όπου υπάρχουν τέτοιου είδου οι περισσότερε περιπτώσει, όπω τη είπα, δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα. Και έχω την εντύπωση, αν τώρα στο Συμβούλιο και εδώ και στο Κοινοβούλιο δεν υπάρχει μια σαφής αντιπαράθεση που θα διεξαρθεί από αυτού, τότε δεν θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ένα πράγμα και να ρωτήσω κάτι. Πρόσφατα υπήρχε μια περίπτωση, μια ιστοσελίδα ε, παιδική πορνογραφία.com λέει. Επρόκειτο για μια σελίδα που ήταν κατά της κακοποίησης παιδιών στην Ολλανδία όμως ε, επευλήθησαν φραγές ε, και παρακολύθηκε και μετά από ένα χρονικό διάστημα επανελήφθη αυτό και είναι ε, αυτή η πορεία με τέτοιου είδους φραγές. Στο τέλος τέλος δεν είναι πραγματικά προβληματικό να επιβάλλονται τέτοιες διαργασίες όταν βρίσκεται υπό εξέλιξη μια νομική προσφυγή. Ο, ο, κύριος Μέλντερ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη ερώτηση προς τον Υπουργό. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ κάτι το Συμβούλιο. Να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που μας είπε. Άλλοι συνάδελφοι. Η κυρία Ήπερ. Ευχαριστώ. Η γερμανική συζήτηση είχε εστιαστεί στην, στο μπλοκάρισμα και στη διαγραφή και δεν θέλω να επεκταθώ διότι είδαμε πόσο σοβαρά θέματα υπάρχουν στην ε, οδηγία αυτή ε, πέραν ε, της κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών. Πρόκειται για θέματα τα οποία άπτονται του αστικού και του ποινικού δικαίου και της προστασίας των παιδιών και γι' αυτό πιστεύω ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλα θέματα πέραν του ότι αναφέρεται εις ε, την ε, ε, οδηγία αυτή και γι' αυτό πρέπει να πω ότι αναφέρουμε σε ένα θέμα που είχε θυγεί από καιρό δηλαδή ότι η οδηγία αυτή δεν είναι συνεπής σε ένα άρθρο μιλάμε για ενός είδους κυρώσεις μετά για άλλου είδους κυρώσεις μετά μιλάμε για κυρώσεις ε, για τα άτομα τα οποία ακόμη δεν έχουν φτάσει ε, στην ηλικία της αυτοδιαθέσεως μετά ε, για κυρώσεις στα άτομα μέχρι 18 ετών δηλαδή ελπίζω ότι με τη συζήτηση αυτή θα μπορέσουμε σε συντονισμό με τις συζητήσεις σε άλλα μέρη να καταλήξουμε σε μια κοινή αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Όχι. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Πρώτα απ' όλα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είπε στην αξιολόγηση της αντιτρομοκρατικής δράσης δεν έχει νόημα η φραγή τέτοιων ιστοσελίδων. Ρωτάω λοιπόν ε, γιατί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν τονίζουμε περισσότερο το θέμα της πρόληψης, εφόσον ξέρουμε ότι το 80% των περοπτώσεων λαμβάνουν χώρα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, οι θύτες είναι άνθρωποι του έμπιστου περιβάλλον του παιδιού. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα για το διαδίκτυο γίνεται η συζήτηση, και το ξέρω, το βλέπω και εδώ, ότι είναι πολύ λεπτό ζήτημα αυτό. Και στη Γερμανία και αλλού γίνονται πολλές συζητήσεις για το πόσο αποτελεσματικό θα ήταν ένα τέτοιο μέτρο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τεράστια συζήτηση, αλλά άμα ξέρουμε ότι τεχνικά είναι εύκολο, μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή ισορροπία ώστε και αποτελεσματικοί να είμαστε και να μην ε, δυσκολεύσουμε τα πράγματα που δεν πρέπει να δυσκολεύσουμε. Η συζήτηση να ξέρετε ότι γίνεται και στο Συμβούλιο. Θα συζητηθεί το θέμα σίγουρα πολύ και το Δεκέμβριο. Δεύτερον, ε, όταν παραγράφεται μια πράξη. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο σημείο αυτό και στο Βέλγιο. Γι' αυτό και γίνεται η συζήτηση και γι' αυτό το θέμα. Ξέρετε, στο Βέλγιο έχουμε και τις περιπτώσεις ε, με την εκκλησία, με τις ε, σεξουαλικές κακοποίησεις παιδιών. Ε, μερικές φορές από κληρικούς και γι' αυτό συζητείται πολύ το θέμα αυτό της παραγραφής. Αυτή ακριβώ είναι η συζήτηση που γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έρχεται και ξανάρχεται. Δεν υπάρχει απόφαση ακόμα. Σίγουρα συμφωνώ για το ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο την πρόληψη. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι Ξέροντας αυτό που είπατε, ότι είναι συνήθως στον κύκλο εμπιστοσύνη της οικογένειας που διαπιστώνονται σεξουαλικές κακοποίησεις, και στο Βέλγιο το είδαμε, Μαθαίνουμε όμως όσο περνάει ο καιρός, ακούμε καινούριε περιπτώσεις, οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε κάποια μέτρα για την ε, πρόληψη παιδαγωγικού χαρακτήρα. Δηλαδή, να φροντίσουμε όλες οι υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με το παιδί να είναι πολύ πιο έτοιμες και προετοιμασμένες να εντοπίσουν κάθε, κάθε είδους υποψία για τέτοιες περιπτώσεις. Όλα αυτά πάντως αποτελούν μέρος Τη συζήτηση που γίνεται στο Συμβούλιο αυτή την εποχή. Θα συζητηθούν το Δεκέμβριο, όπως σας είπα, και τότε περιμένουμε να υπάρξει κάποια απόφαση. Και για τα θέματα στα οποία δίνετε εσείς προτεραιότητα. Ελπίζω τον Ιανουάριο να μπορέσουμε να έχουμε μια τελική απόφαση. Ελπίζω να γίνει αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα και να έχουμε προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα πριν την Ουγγρική Προεδρία. Η συγκίτρια δεν λέει ότι θέλει να επανέλθει. Θέλει ή όχι. Όχι. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Συνάδελφοι, ερχόμαστε έτσι στο σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως και με συγχωρείτε που σας πιέζω, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής οδηγίας 2003-109-ΕΚ ε, στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η συγητής Νοκλόντ Μοράς, ποιος, ε, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τώρα τα αποτελέσματα της, ε, τρίτης, ε, τρι, της δεύτερης τριμερούς διαπραγματεύσεως στις αρχές Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Ίσως ορισμένοι συνάδελφοι δεν ήξεραν ότι σε κάποιο σημείο δεν θα είχαμε διερμηνία και σας ευχαριστώ που επιταχύνατε. Έχουμε φτάσει στον τριμερή διάλογο έχοντας διευκρινίσει τα διάφορα θέματα και τα οποία θέλουν μελέτη και γι' αυτό θα αναφερθώ στους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι με στήριξαν και με βοήθησαν στο θέμα αυτό. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο όπου έγινε ο τελικός τριμερής διάλογος ε, με ορισμένα θέματα που έπρεπε να επιληθούν. Καταρχήν, πόσο, πώς θα υπολογιζόταν η περίοδος ετήσεως, ετήσεως ε, ε, ασύλου σε σχέση με την διαμονή και καταλήξαμε σε μία συμβιβαστική λύση 18 μηνών μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ευχαριστώ και τις δύο πλευρές που μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτό το συμβιβασμό και ε, ένα άλλο θέμα που δεν είναι θέμα της Επιτροπής μας ή της εκθέσεως αυτής αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο το κοινοβούλιο, δηλαδή τον πίνακα συσχετισμών. Διότι είχαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με τον πίνακα συσχετισμών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως θα θελήσει να, σχολιάσει, να σχολιάσει το θέμα αυτό, διότι πίστευαν ότι μπόρεσαν να κάνουν κάποια εξαίρεση παρόλο που δεν έχουν υποχωρήσει στο ότι χρειάζεται να υπάρχουν οι πίνακες συσχετισμών σε όλες τις εκθέσεις για να εξασφαλιστεί η σωστή ποιότητα εφαρμογή στην εθνική νομοθεσία αυτών των νομοθετημάτων και όσον αφορά το τελικό θέμα, ε, χαίρομαι ότι επιτύχαμε ε, διότι καταλήξαμε σε μία βάση ε, με την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε. Μόνο ο Αλεξάνδρ Αλβάλο βλέπω να ζητά το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη σας είπα ότι αν χρειαστεί να πάρω το λόγο ε, και πάλι το πράτο εν ονόματι της Σεσίλια Βίκστρεμ που ήταν ισχυώδη στον τομέα αυτό και η οποία λέγει ότι ήταν ε, μεγάλη, μεγάλο επίτευγμα που καταφέραμε να έχουμε μία κατάληξη σχετικά με το άσυλο και ελπίζουμε θα καταλήξουμε ε, επίσης σε καλή έκβαση και σε άλλα θέματα. Βεβαίως όσον αφορά τους ε, πίνακες συσχετισμών για να υπάρξουν συμφωνίες ε, πρέπει να πούμε ότι σε ορισμένους ε, τομείς είναι ανησυχητική εξέλιξη αυτή ιδίω όσο αναφέρεται ή στη Συμφωνία Δουβλίνο 2 επί της οποίας είναι η συγγήτρια η Σεσίλια και ας ελπίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει υπόψη της αυτά τα στοιχεία όταν θα προχωρήσει και επίσης ε, συγχαίρει το Κοινοβούλιο που μπόρεσε να ολοκληρώσει το θέμα αυτό με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος ζητά το λόγο, όχι. Ωραία. Τότε θα δω αν υπάρχει εδώ κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος ενδεχομένως θα ήθελε να σχολιάσει. Δεν βλέπω να υπάρχει κανείς. Υπάρχει. Α, μάλιστα. Η κυρία Γκιάν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλώς θέλω να σας πω ότι και εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Να ευχαριστήσω δηλαδή τον εισηγητή κύριο Μωράη σχετικά με, αυτή την, ε, με αυτό το φάκελο και να διευκρινίσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον πίνακα συσχετισμών διότι ο φάκελος αυτός είναι πολύ σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό δεχτήκαμε να υποχωρήσουμε σχετικά με τον φάκελο αυτό τελείως εξαιρετικά για να ε, δώσουμε ένα θετικό σήμα για την προώθηση ορισμένων μέτρων για το πρόγραμμα του ασύλου και επιπλέον ε, να μπορέσουμε ε, να προσεγγίσουμε το Συμβούλιο επί του θέματος αυτού ελπίζοντας ότι και τα άλλα θεσμικά όργανα θα συνεχίσουν να συζητήσουν συζητούν ε, τα θέματα αυτά και άλλωστε θα διατυπώσουμε μία δήλωση επί του θέματος. Ευχαριστώ. Κλοντ, έχεις κάτι άλλο να πεις? και προς τον ε, Αλεξάνδρε για τους φιλελεύθερους και τους φίλους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να τονίσω ότι η κατάσταση έχει ως εξής. Εμείς επιμένουμε στη θέση μας για τον πίνακα συσχετισμών αφενός και δεύτερον η βασική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να προωθήσει το πακέτο του ασύλου και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για το Κοινοβούλιο φτάνοντας στις επόμενες φάσεις του πακέτου του ασύλου και αυτός είναι ένας ουσιαστικός λόγος για τον οποίο προχώρησε το πακέτο αυτό. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, αλλά με, με διέκοψαν και πρέπει να ξαναοργανώσουμε την ε, ημερήσια διάταξη. Άρα με αυτό ολοκληρώσαμε το σημείο 6, τη συζήτησή του. Έχουμε ακόμη πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα έλεγα ότι το τελευταίο θέμα σχετικά με την οδηγία εναντίον των διακρίσεων να μεταφερθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Οπότε έχουμε μία ώρα για τα υπόλοιπα θέματα, εκ των οποίων δύο είναι παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Νακροτικών που έπρεπε να ξεκινήσουν στις 4.30. Ε, Δεν νομίζω θα μπορέσουμε να κάνουμε 15 λεπτά δύο συζητήσεις αλλά τώρα έχουμε τις ελάχιστες απαιτήσει για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας αναδιατύπωσης. Θα σας δώσω το λόγο και μπορείτε να μου πείτε τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι διότι οι σκιώδεις στο σημείο αυτό μπόρεσαν να έχουν μία πολύ εκτεταμένη συνεδρία στην περασμένη εβδομάδα με διερμηνία για να εξετάσουν τις τροπολογίες διότι δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε περίπου 100 τροπολογίες σήμερα. Ίσως θυμάστε ότι ήταν ε, μία ε, ε, ε, ε, μία ενημέρωση όσον αφορά την διατύπωση του προγράμματος της Στοχόλμης και ακόμη και η γαλλική και η γερμανική ε, κυβέρνηση είπαν ότι ήθελαν να υπάρξει μία ε, ε, ακριβή συμμόρφωση στο ε, έγγραφό τους. Λοιπόν, κοίταξα την αρχική μου έκθεση για την αναδιατύπωση και τώρα θα δείτε ότι είχαμε πολλές τροπολογίες και από άτομα και από πολιτικές ομάδες και καταλήγουμε σε κάπου 100 τροπολογίες. Ελπίζαμε ότι θα είχαμε ε, ε, ευρεία συνένεση σε διάφορα θέματα και να υποφεληθούμε από τη Βελγική Προεδρία που τουλάχιστον ήθελε να συζητήσει το θέμα μαζί μας αλλά με τον αριθμό των τροπολογιών και με τις διαφορετικές απόψεις από τις οποίες αποκλίνουν οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δικές μας δεν βλέπω να προχωρέσουμε βάσει του χρονοδιαγράμματος εγκαίρως διότι πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες δεν θέλουν να μελετήσουν τις τροπολογίες και ε, να προχωρήσουν σε ένα πιο οργανωμένο σύστημα. Ε, προβλέπω λοιπόν ότι θα ξανασυζητηθεί στην Επιτροπή τέλος Νοεμβρίου. Δεν νομίζω όμως, αλλά γιατί δεν νομίζω ότι θα έχουν ε, όλοι καιρό να το κοιτάξουν. Άρα προτιμάτε ίσως να μην συζητήσουμε ε, και να μην ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στις 9 Δεκεμβρίου πριν από το τελευταίο Στρασβούργο του έτους. Οπότε κατόπιν αυτού η επόμενη δυνατότητα ψηφοφορία πορεία στην Επιτροπή θα είναι στι αρχές του χρόνου υπό Ουγγρική Προεδρία όπου τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Ε, όσον αφορά τις τροπολογίες. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες οι οποίες είναι εκτός ε, της ε, εμβέλειας της αναδιατυπώσεως. Δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε με την Επιτροπή με αυτά τα θέματα και ε, μόνο θα προχωρήσουμε μόνο στα θέματα όπου υπάρχει ευρεία συνένεση αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τα υπόλοιπα διότι πολλά αναφέρονται ή στην αναδιατύπωση και στην μορφή της οδηγίας και είναι ως τούτου σημαντική, σημαντικές. Βλέποντας απλώς όμως τον, τίτλο της αναδιατύπωσης την, ε, το διαχωρισμό σε δύο κατηγορίες ε, την διατύπωση για την ανθρωπιστική βοήθεια η οποία είναι μία ομπρέλα μεταξύ ε, των δύο ειδών προστασίας ουσιαστικής και δευτερογενής ή επικουρικής θα ήθελα να σας πω ότι αρχίζω να ε, αγχώνομαι με το όλο θέμα και γι' αυτό θα πρέπει να ετοιμάσω ένα σημείωμα με μία ανάλυση των διαφόρων ε, θεμάτων που διακυβεύονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν όλοι να ε, έχουν μπροστά τους ένα χαρτί στο οποίο να μπορούν να αναφέρονται αντί να ψάχνονται μεταξύ 100 τροπολογιών. Ε, ευχαριστώ. έχω τρεις υποψηφίους ομιλητές, αλλά εάν η ψηφοφορία μένει για τον Ιανουάριο Ίσως θα βρούμε κάποια στιγμή για να συζητήσουμε εκτενώς το θέμα αυτό κάποια άλλη στιγμή και όχι από τώρα στον Ιανουάριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τότε πάλι ενωνώ με ε, της κυρίας ε, Μέτια Χέρση η οποία ε, δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και εφόσον θα συζητηθεί κάποια άλλη τιμή, στιγμή θα ήθελα απλούστατα να υπενθυμίσω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας καθορισμός στον όρο, δηλαδή της οδηγίας και όλων των σχετικών θεμάτων και ε, ποια είναι η θέση η οποία να δίδεται εις τους πρόσφυγες είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε με τον, την εισηγήτρια γνωρίζετε τις θέσεις της κυρίας Χάρστ και ίσως για να παραμείνω πολύ σύντομος εφόσον έχω ήδη μιλήσει προηγουμένως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να δούμε αν είναι ε, ε, σκόπιμο να ανοίξουμε την αγορά εργασία στους πρόσφυγες για να μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύω όμως ότι θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε περισσότερο στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ για τη σύντομη παρουσία σας κυρία Χολμάγερ. Ε, κυρία Πρόεδρο, οι αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη ε, και ε, θέλω να ευχαριστήσω την Τζιν Λάμπερτς για τη συνάντηση που είχαμε ε, και ε, μπορέσαμε να διευκρινίσουμε πολλά θέματα τα οποία ακόμη θέταμε μεταξύ μας, δηλαδή νομικές διευκρινήσεις οι οποίες ήταν αναγκαίες για το θέμα της υπηκοότητος ή για τη δυσκολία της, του διαχωρισμού μεταξύ των προσφύγων και των επικουρικώς προστατευομένων ατόμων και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε εφόσον έχουμε χρόνο να ξανασυναντηθούμε και να διευκρινίσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ακόμη πράγμα το οποίο έθιξε η Σιλβίγκη Γιόμ δηλαδή την τροπολογία 34, τροπολογία 34 όπου Ήθελα να ρωτήσω ε, μέχρι ποιο σημείο προβλέπετε ότι στο μέλλον ε, δεν ε, θα διατυπώνουμε για τον όρο «απατρίς» αλλά θα είναι ετούντες οι οποίοι ε, κάνουν μία αίτηση εντός μίας χώρας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή ε, ε, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι και ένας Ευρωπαίος πολίτης, ένας Ρουμάνος στη Γαλλία ή ένας Γάλλος στην Αγγλία. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι η σκοπιμότητα αυτής της τροπολογίας εφόσον ε, θα έπρεπε να μας το εξηγήσετε αυτό για να δούμε τι καλύπτεται πίσω από, αυτήν, την, ε, αυτό το θέμα. Με συγχωρείτε που είμαι ε, τόσο βία, αλλά ε, ε, αντιλαμβάνομαι ότι με την ταχύτητα αυτή δεν προλαβαίνουν να μεταφράσουν. Αν λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε περαιτέρω, υπάρχουν, μπορούμε να συζητήσουμε μετά τις 5 και 4 χωρίς διερμηνία, αλλά πολλοί θα παραπονεθούν, γι' αυτό και προσπαθώ να τα, όλα αυτά να τα συγκεράσω. κυρία Ρωμέρο Λόπες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Τζιν Λάμπερτς για τη δουλειά της και για τις τροπολογίες που υποβάλλει στο κείμενο. Χαίρομαι που τελικά υπήρξε προσέγγιση. Αυτό που είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου στην οδηγία αυτή είναι να πετύχουμε το ανώτατο δυνατό επίπεδο συμφωνίας. Για την τροπολογία Σιλβίκη Γιώμ δεν μπορώ να σχολιάσω. Εκείνη το ζήτησε είναι πάντως μία τροπολογία που εδώ και καιρό ζητούν διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλά πρέπει να δούμε νομικά κατά πόσο στέκει. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο σε βάθος την τροπολογία αυτή. Τίποτα άλλο, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Όπως είπε πάντως και η κυρία Λάμπερτ, αξίζει μια συζήτηση περισσότερο σε βάθος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιακολίνο, ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και συγγνώμη. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή όσα είπαν η συγγήτρια και όσοι πήραν το λόγο μετά. Πιστεύω ότι, ένα... ότι το κείμενο είναι καλό. Πρέπει όμως να επαληθεύσουμε ποιες είναι ακριβώς οι προϋποθέσεις εκείνες που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε με αυτή την πρόταση. Αλλιώς κινδυνεύουμε να έχουμε ετοιμάσει κάτι το οποίο τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν όσον αφορά τους ανήλικες για παράδειγμα. Και εδώ πρέπει να υπάρξουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Όταν θα έχουμε αξιολογήσει και το καθεστώ τους και την αντικειμενική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, τότε θα πρέπει να αγγιόμεθα κάθε είδους βοήθεια, υγεία και οτιδήποτε άλλο στους δικαιούχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος στο κατάλογο μιλητών. Παρακαλώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Τζιν Ελπίζω με τις τροπολογίες να δούμε και το θέμα της δίωξης ατόμων, τα οποία ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή θεωρούν κάποιοι άλλοι ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα, σε μια εθνική μειονότητα ή βρίσκονται δίπλα και κάποιοι νομίζουν ότι ανήκουν σε αυτή την εθνική μειονότητα. Μπορεί να είναι πρόβλημα αν μπουν στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Ποιοι θα το είπατε ότι ε, διώκεστε επειδή ανήκετε στη συγκεκριμένη εθνική μειονότητα, αλλά δεν ανήκετε τελικά σε αυτήν. Θέλουμε λοιπόν να συμπεριλάβουμε σε μια τροπολογία και τις δύο περιπτώσεις, γιατί στο κοσυφοπέδιο δεν έχει σημασία αν είναι πραγματικά μερικές φορές από μια συγκεκριμένη εθνική μειονότητα ή αν ε, υπάρχει αντίληψη ότι ανήκουν σε αυτήν την εθνική μειονότητα. Το θέμα είναι ότι διώκονται. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε, δεν έχει στήσει κανένα άλλο το λόγο, λέει η πρόεδρος ή η συγκήτρια τώρα, η κυρία Λάμπερτ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέρφους για αυτά που είπαν και το ενδιαφέρον του. Όπως είπα θα ετοιμάσω λεπτομερώς της και θα μπορέσουμε να δούμε και την 34 για να δούμε ακριβώς ποια είναι. Τόσο μπορεί να μην είναι 34. Λυπάμαι που συζήτησα τόσο σύντομη σήμερα. Θα επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και ζητώ και εγώ συγγνώμη, αλλά προσπαθώ να απολέψω τα πράγματα. Τώρα. Η μέρη συνέταξη προβλέπει τώρα παρουσίαση της ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Δεν τον βλέπω όμως εδώ. Okay. As he's not here and the... Δεν είναι εδώ. Η παρουσίαση για τα ναρκωτικά προβλέπεται αργότερα, οπότε θα περάσουμε τώρα στην έκθεση του κύριου Μπουσέτελ, που μόλις σας μοιράστηκε μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε λίγο χρόνο για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εναλλακτική λύση είναι να το αναβάλουμε και να συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά τότε θα είναι πέμπτη απόγευμα, οπότε και αυτό είναι το ιδεώδες. Οπότε ας ξεκινήσουμε και βλέπουμε πώς θα προλάβουμε να προχωρήσουμε. Μπουσάτιλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζω σήμερα στους συναδέλφους την έκθεση που εγώ ετοίμησα όσον, ε, ετοίμασα όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την Frontex. Πρόκειται για τον συντονισμό της συνεργασίας των κρατών μελών σε θέματα εξωτερικών συνόρων. Έχουν ήδη γίνει διάφορες συναντήσεις με την Επιτροπή, με το Συμβούλιο, με την ίδια τη Frontex, την οποία και επισκέφθηκα σήμερα πριν έρθω εδώ. Είχαμε και συναντήσεις με τους κοιόδες εισηγητές, αλλά και με εκπροσώπους του ΙΠΙΕΣ και όλους τους ενδιαφερόμενους. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων εδώ, σε αυτή την Επιτροπή. Η έκθεση που έχετε σήμερα μπροστά σας περιλαμβάνει 68 τροπολογίες θα τις χώριζα σε 10 διαφορετικές κατηγορίες για 10 διαφορετικά σημεία. Μια που μας κάνετε να βιαζόμαστε τόσο πολύ σήμερα κυρία Πρόεδρε, θα αναφερθώ στα 5 εγώ θέματα. 5 από τα 10 σημεία στα οποία υποβάλλω τροπολογίες. Πρώτον, η έκθεση θέλει να ενισχύσει τόσο αναφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους συναδέρφους από άλλες πολιτικές ομάδες επίσης. Δεύτερον, προτείνω σε όλους τους συναριοφύλακες που συμμετέχουν ε, σε δράσεις της Frontex, είτε πρόκειται για μικτές, είτε πρόκειται για το Rapid Border Intervention, τέτοιες αποστολές, και στις δύο περιπτώσεις να τους ονομάζουμε βάσει αυτού που πραγματικά είναι. Δηλαδή, συνοριοφύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό είναι. Έτσι να ονομάζονται. Τίποτα άλλο. Προτείνω λοιπόν αυτή την αλλαγή. Τρίτον, προτείνω η Frontex να έχει ένα ρόλο όχι μόνο ε, θέση εφαρμογή των ε, επιστροφών, των υποχρεωτικών, αλλά και των σε θελοντική βάση. Τέταρτον, προτείνω ο οργανισμός να έχει ως αρμοδιότητα να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μόνο έτσι μπορεί να φέρει σε πέρα στα καθήκοντά της. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα αυτό και ακριβώ γι' αυτό προτείνω αυτό να γίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Τέλος, θέλω να αυξήσω το δημοκρατικό έλεγχο του οργανισμού, επιτρέποντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μεγαλύτερο ακόμα ρόλο στον έλεγχο της δουλειάς του οργανισμού και ιδιαίτερα όταν πρόκειται και για τρίτες χώρες. Αυτές είναι οι κυριότερες πέντε αλλαγές από τις δέκα που συνολικά προτείνω στην έκθεση αυτή. Από εκεί και πέρα περιμένω αντιδράσεις των συναδέρφων και τροπολογίες τους. Θέλω επίσης να πετύχω ευρεία συνένεση πάνω στο κείμενό μου. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ που ήσασταν και συνεργάσιμος. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Ας τους ακούσουμε πρώτα και μετά η Επιτροπή και το Συμβούλιο που μπήκαν τελευταία στιγμή θα προλάβουν να ηρεμήσουν λίγο και να είναι έτοιμοι να μας απαντήσουν. Ε, λοιπόν, Άλβαρο και Κέλλερ. Άλβαρο, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και σε εσάς Πρόεδρε, και στον εισηγητή που 120 λεπτά ημερήσιας διάταξης εσείς μπορέσατε και τα βάλατε σε 60 λεπτά. Για την έκθεση Frontex τώρα και για τον Σάιμον. Σε ευχαριστώ πολύ από τους σκιώδες μας εισηγητές για την καλή συνεργασία που έχεις μαζί τους. Η Σεσίλια Συμφωνεί απόλυτα μαζί σου για την ξεκάθαρη εντολή και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης λέει ότι τα λαμβάνει υπόψη σου. Αναφέρθηκε στις τρίτες χώρες, στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, για τα προσωπικά δεδομένα επίσης κάτι είπες. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η διαδικασία αυτή, επεξεργασία δηλαδή προσωπικό δεδομένο, πρέπει να είναι σε περιορισμένο βαθμό. Αυτό που δεν είπες είναι για τον εξοπλισμό της Frontex και για το κόστος. Ότι θα μπορούσαμε ίσως να τον δανειζόμαστε αυτόν τον εξοπλισμό. Πρέπει να δούμε πόσο κοστίζει σε αυτή την περίπτωση, μήπως είναι πιο λογικό από την αγορά. Ελπίζω να πετύχουμε συμφωνία, που δικιά μας την πλευρά θα υπάρξει. Κατά τα άλλα, καλή τύχη και άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Πρόεδρε, συγχαρητήρια και σε εσά πάλι. Όταν παίρνετε φόρα, είναι δύσκολο να τα βγάλει κανεί μαζί σα. Είσαστε όμω αποτελεσματικοί παρόλα αυτά. Μπράβο. Ευχαριστώ. Συνήθω δεν είμαι έτσι, δεν παίρνω φόρα, είμαι πιο ήπια. Η κυρία Κέλλερ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή συνεργασία που είχε με του σκιώδει εισηγητέ. Ε, δεν έχω δει και τι 50 τόσε σελίδε στα 5 λεφτά που μου έχει μοιραστεί το κείμενο. Αυτό που συγκρατώ πάντω από την παρουσίασή σα είναι κάποια καλά θέματα. Ενίσχυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα. Περιμένω φυσικά τις λεπτομέρειε. Δημοκρατικός έλεγχος και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, ζωτική σημασία. Μπράβο. Για τα προσωπικά δεδομένα, ίσως να έχουμε διαφορετική άποψη. Όπως φαντάζεστε. Θα υπάρξουν κάποιε τροπολογίε από την πλευρά μα αναφίβολα. Αλλά πιστεύω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Μπρόντς, επόμενος ομιλητής. Λοιπόν, ε, εκπλήσωμε διότι αμφισβητούμε τα προσωπικά δεδομένα, διότι διαφορετικά πώς θα προστατεύαμε τα σύνορα της Ευρώπης. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, αλλά πιστεύω ότι οι προσπάθειές τους υποθάλπονται μέσω των προσπαθειών των ατόμων να ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες, να μπαίνουν από την κυρία είσοδο, ενώ τους εμποδίζουν να μπαίνουν από το πλάι. Λοιπόν, ε, Τώρα θα ήθελα να σχολιάσει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστώ. δεν ήρθαμε αεροπορικός, οπότε ήρθαμε γρήγορα. Πρέπει όμως να σας πω ότι θα είμαι πάρα πολύ σύντομος διότι μόλις λάβαμε το έγγραφο αυτό οπότε δεν είχαμε ακόμη χρόνο να το εξετάσουμε και ατυχώς ε, δεν άκουσα την παρουσίαση της εισηγήτριας, οπότε προς το παρόν επιφυλάσσουμε τη θέση μας. Ε, έτσι βέβαια μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι αντιθέτως το ότι είπατε το Συμβούλιο δεν έχει έρθει ακόμη. Δηλαδή ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου δεν είναι εδώ. Α, είναι εδώ αλλά δεν έχει μιλήσει. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του Συμβουλίου αλλά δεν μπορεί να παρέμβει, άρα ξαναδίνουν το λόγο στον κύριο Μπουσουτήλ, τον εισηγητή. Ε, είναι κατανοητό διότι μόλις ε, ε, παρουσιάσαμε αυτήν την έκθεση και θα ήθελα να απαντήσω στον Αλεξάνδερ Άλβαρο για τις παρατηρήσεις του, διότι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσουμε την δυνατότητα να έχουμε το δικό μας εξοπλισμό ε, είναι ένα νέο θέμα γιατί δεν είναι ε, μόνο κάτι το οποίο έχω προτείνει αλλά και το οποίο στηρίζω σαν εγχείρημα. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι προσλέπω εις ε, τα σχόλια όλων των ενδιαφερομένων και των δύο άλλων θεσμικών οργάνων και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε, έναν ευρύτατο, σε μια ευρύτατη συνένεση σχετικά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι την 3η 14 μεσημέρι και θα συζητηθεί στις 25 και 26 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Ελευθεριών. Και φτάνουμε τώρα στο επόμενο θέμα και θα έλεγα να ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση της ε, ε, ετήσιας ε, εκθέσεως για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το 2010. Θεωρώ όμως ότι είναι πρόωρο να παρουσιάζεται η έκθεση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω ε, τον ε, Διευθυντή του Κέντρου να μας το παρουσιάσει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη διερμηνία μέχρι τις 5 ε, παρατέταρτο και τέταρτο, οπότε θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι διότι όπως κάθε χρόνια σας παρουσιάζω τα βασικότερα θέματα της ετησίας εκθέσεώς μας τώρα για το 2010 σχετικά με τα προβλήματα ναρκωτικών και τοξικομανίας. Βεβαίως εφέτος θα μπορούσαμε πολύ απλά να πούμε ότι ε, η ε, κατανάλωση ναρκωτικών ε, είναι σταθερή στην Ευρώπη αλλά θα είχαμε παραβλέψει ότι γίνεται πολύ πιο ε, περίπλοκη η κατανάλωση αυτή και ότι έχουμε να κάνουμε με, ένα, πιο, με μια πιο περίπλοκη αγορά από ό,τι στο παρελθόν και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη εις την επόμενη στρατηγική μας, δηλαδή για το 2013 έως 2020. Όσον αφορά τις ε, ε, ε, τις λεπτομέρειες θα ξεκινήσω με την ηρωίνη. Η ηρωίνη που είναι το μεγαλύτερο πλήγμα για την Ευρώπη διότι τα περισσότερα θύματα είναι καταναλωτές της ηρωίνης και έχουμε 7-8 χιλιάδες θανάτους που οφείλονται ε, σε κατάχρηση αυτού του ναρκωτικού πλέον. Έχουμε δύο έως 3.000 τοξικομανής ε, της ηρωίνης τα τελευταία χρόνια και αυτό διότι τα τελευταία χρόνια η ε, καλλιέργεια αυτών των οπιοειδών στο Πακιστάν έχει αυξηθεί. Η χειρότερη και πιο βλαβερή μορφή βέβαια είναι η κατανάλωση ηρωίνης υπό μορφή ενέσιμη και γι' αυτό προσπαθήσαμε ε, για για τοξικομανείς όπου υπάρχει ε, τα βίβαση ασθενειών όπως το AIDS να ε, παρέμβουμε και να μειώσουμε αυτή την, ε, αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που μας να ανησυχεί είναι η τεράστια τοξικομανία η την Ρωσία και στην Ουκρανία και η κατάσταση στις δύο αυτές χώρες πρέπει να εξεταστεί και χρήζει της βοηθείας μας διότι όταν μιλάμε για άλλες ουσίες η ε, ε, κοκαίνη, οι αμφετεμίνες και η έκσταση παίζουν βασικό ρόλο στην Ευρώπη διότι έχει αυξηθεί η ε, κατανάλωση κοκαίνης πολύ και αυτή τη στιγμή είναι η, πολύ, δεύτερη πιο πολύ πολύ καταναλωνόμενη ουσία στην Ευρώπη. Ε, η υψηλή κατανάλωση της ε, κοκαίνης υπάρχει ε, σε λίγες χώρες αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες αυξάνεται και αυξάνεται ιδίως στις πιο εύκολες, εύπορες κοινωνικές τάξεις πράγμα το οποίο οδηγεί σε ανάγκη ε, θεραπείας, σε αύξηση των θανάτων και σε κόστος για την κοινωνία. Η ε, πρόοδος όμως της κοκαίνης δεν εμφανίζεται μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρική και στην Ασία ε, διότι το εμπόριο οδηγεί σε μία αποσταθεροποίηση αυτών των περιεχών και επιπλέον ως αντίδραση εις τις κινήσεις των διοκτικών αρχών ιδίως στην Ιβηρική Χερσόνιο ε, έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές ε, ε, αγορές ή στην Βόρειο Αφρική. Πέραν αυτού όμως υπάρχει πολύ υψηλή κατανάλωση αμφεταμινών στην Ευρώπη και η έκσταση παίζει μεγάλο ρόλο διότι θεωρούμε ότι η ουσία αυτή έχει καταναλωθεί από 2,5 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη πέρυσι. Ε, υπάρχουν ουσίες όπως η BCP ή η μεθετρων που πουλούνται στην αγορά και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ε, δεν έχουν αποδώσει διότι οι έμποροι τα παρακάμπτουν. Για πολλούς νέους λοιπόν η, κατανάλωση μειγμάτων έχει αυξηθεί από τους νέους. Ε, δεν μπορώ ε, λόγω του περιορισμένου χρόνου να επεκταθώ στο θέμα των βλαβερών συνεπειών της ε, καταναλώσεως τοξικών ουσιών ιδίως με συνδυασμό νοπνευματοδών παρόλο που οι νέοι έχουν καταλάβει εντωμεταξύ το μήνυμα που έχουμε απευθύνει στο θέμα αυτό. Αλλά όσον αφορά τώρα η, την ε, κάναβη ε, χρησιμοποιείται ε, πέρυσι κατανάλωσαν 23 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ε, καναβή και 75 εκατομμύρια την έχουν δοκιμάσει κάποια στιγμή. Η αξιολόγηση των βλαβών που προκαλεί η κάναβης δεν είναι εύκολη, αλλά πολλοί νέοι την, εγκαταλείπουν την ουσία αυτή προτού τους προκαλέσει σοβαρές βλάβες και ε, δεν ε, σημειώνουμε πολλά παραδείγματα αναπνευστικών ασθενειών παρά μόνο πολλά χρόνια μετά ε, και γι' αυτό η σχέση μεταξύ των, της χρήσεως ε, κανάβεως και ε, ψυχοσωματικών ασθενειών ε, πιστώνεται όλο και περισσότερο. Υπάρχει μια συνεχής αύξηση της Ευρώπης. Βλέπω ότι υπάρχει και μεγά, σημειώνω ότι υπάρχει και μεγάλη καλλιέργεια της κάναβης σε συνεργασία με την οργανωμένη εγκληματικότητα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να συνδυάσει το εμπόριο ναρκωτικών με την κάναβη και αυτό αποτελεί ένα ε, ακόμη παράδειγμα των εξελίξεων εις ε, την αγορά ναρκωτικών. Υπάρχουν και ε, εργαστήρια για την διήλυση των ναρκωτικών, παραδείγματος χάρη για την βελτίωση της κοκαίνης η οποία έχει εισαχθεί παρανόμως. Ε, έχουμε επίσης με την Ευρωπόλο ε, μία υπηρεσία για ένα σύστημα έγκαιρης ενημερώσεως για νέα ναρκωτικά και έχουμε σημειώσει 24 νέα, ε, νέες, νέες τέτοιες ουσίες και για του χρόνου θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων νέων ουσιών Λοιπόν, όπως ε, οι κατινόνες ε, οι οποίες είναι μια εναλλακτική λύση για την έκσταση ή την κοκαίνη. Ε, έχουμε ήδη έναν αριθμό θανάτων και υψηλή κατανάλωση αυτών των ουσιών και γι' αυτό έχει γίνει μία μελέτη αξιολογήσεως των επιπτώσεων και υπάρχει απαγόρευση χρήσεως της ουσίας αυτής εντός των επομένων εβδομάδων θα προχωρήσει και η απόφαση από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών, ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά τα συνθετικά καναβοειδή ε, που παράγονται από την ουσία TAC ε, έχουν, ε, ε, έχουν εντοπιστεί από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και προσπαθούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ε, τα μέτρα ελέγχου έχουν όμως επιτύχει και δεν είναι πλέον εύκολο να απολυθούν οι ουσίες αυτές, τα μείγματα αυτά μέσω του διαδικτύου και προσπαθούμε να ελέγξουμε τις πωλήσει μου αρέσει διότι ε, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους ε, δυνητικούς καταναλωτές για τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται η κατανάλωση αυτών των ουσιών. Ε, είναι δύσκολη η ενημέρωση αυτή διότι τα, οι ονομασίες αλλάζουν συνέχεια. Μέχρι στιγμής ξέρουμε 170 καταστήματα online στην Ευρώπη που μπορούν να πωλήσουν σε Ευρωπαίους πολίτες πράγμα το οποίο δείχνει ότι δεν πρέπει κανείς να παρανοεί την εξέλιξη αυτή και για να υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός έλεγχος δεν υπάρχει μία δεδομένη λύση. Ξέρουμε όμως ότι ορισμένες ουσίες είναι πιο βλαβερές από άλλες και γι' αυτό θα πρέπει να ανταλλάσσουμε εμπειρίες στην Ευρώπη για να βελτιώσουμε βελτιώσουμε τις γνώσεις μας. Το θέμα το οποίο με, μου έχει τεθεί τελευταίο στο πιο συχνά από δημοσιογράφους είναι πώς θα επηρεάσει τον τομέα αυτό των ναρκωτικών η οικονομική κρίση. Δηλαδή όποιος έχει, έχει λιγότερα χρήματα θα χρησιμοποιεί λιγότερα ναρκωτικά. Μπορεί όμως να συμφεί και το αντίστροφο. Δηλαδή αν κάποιος χάσει τη δουλειά του θα ξεκινήσει να πειραματίζεται με ναρκωτικά ή να καταναλώνει ε, σε δύσκολες λοιπόν οικονομικές ε, περιόδους επιδεινώνεται η κατάσταση της χρήσης ναρκωτικών και υπάρχει ο κίνδυνος παραδείγματο χάρη να ε, υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες και ε, γι' αυτό εάν περιορίσει κανείς την προσφορά και βελτιώσει την πρόληψη θα μπορούσαμε ε, να ε, έχουμε ενδεχομένως περιθωριοποιήσεις και πολιτικά προβλήματα. Εντάξει, ας μην μιλώσουμε τον προϋπολογισμό αλλά ξέρουμε ότι σε ορισμένα κράτη δεν υπάρχουν δυνατότητες πρέπει να περιοριστούν οι χρηματοδοτήσεις οπότε αν η χρηματοδότηση μειωθεί στον τομέα αυτό και αν είναι απαραίτητο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εις ε, το παρελθόν ε, ορισμένα μέτρα απέδωσαν ενώ άλλα έχουν αποδώσει λιγότερο και πρέπει να μειώσουμε και την εγκληματικότητα των αρκομανών και να βελτιώσουμε την κατάσταση της υγείας τους. Κάνω λοιπόν μία έκκληση. Όταν ε, αποκλείονται οι μειώσεις των χρηματοδοτήσεων τότε θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα κατά των ναρκωτικών κατά προτεραιότητα. Ένα πρακτικό παράδειγμα. Βρίσκονται ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι σε θεραπεία και παίρνουν ένα υποκατάστατο θεραπεία. Τα τελευταία 15 χρόνια η ζήτηση για τη θεραπεία αυτή διαρκώς αυξανόταν και όλο και περισσότεροι ε, οργανισμοί και ε, θεραπευτήρια προσφέρουν αυτή την ε, θεραπεία. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε σταθεροποίηση του αριθμού χρηστών στην Ευρώπη. Και πέρα από αυτό βλέπουμε ότι η ζημιά όσον αφορά τον κοινωνικό περίγυρο μπορεί να ε, μειωθεί. Αλλά έχουμε και άλλα μέτρα παράδειγμα εκστρατείε ε, στα μέσα η, η σύλληψη των καταναλωτών είναι δαπανηρές ε, δυνατότητες αυτές και πολύ λιγότερο ευθύης ε, για την κοινωνία. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι έργο του παρατηρητηρίου για την εξάρτηση είναι στο συνολικό εύρος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ναρκωτικών στην Ευρώπη και να ενημερώνει για τα μέτρα και τις δράσεις. Παρότι είναι υπερβολικά φορτισμένο ένα ένα τέτοιο θέμα και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί αντικειμενικά. Θέλω να πω ότι επιστημονικά και αντικειμενικά πρέπει να εξετάζονται αυτά τα θέματα, διότι μόνο σε στοιχεία βασιζόμενη συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε στοχοθετημένα αποτελεσματικά μέτρα. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και νομίζω είναι θελκτικό ελκυστικό η συζήτηση που έχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωκοινοβούλιο που είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν κάποιοι για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας. Τώρα θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε αυτά και πιεστικά όλας λόγω της κρίσης. Έχουν τρει ζητήσει τον λόγο να περιοριστείτε σε ένα λεπτό καθένας παρακαλώ. Αυστηρά ένα λεπτό η παρέμβασή σας και μετά θα υπάρχει χρόνος για ε, τις απαντήσεις προτού περάσουμε στο επόμενο. Ο κύριος Γιακουλίνο, μετά ο κύριος Μπρόντς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή πρέπει να πω παρακολούθησα τα όσα είπε ο Διευθυντής του Παρατηρητηρίου. Με ιδιαίτερη προσοχή τον άκουσα. Και τούτου λεχθέντος πολύ συγκεκριμένα και χειροπιαστά στοιχεία παρουσίασε και όσον αφορά και τα παλαιότερα κράτη-μέλη. Η ε, πολιτική κατά των ναρκωτικών και η αντιμετώπιση των ναρκωτικών μπορεί κανείς ε, να πει συγκεκριμένα ε, για αυτά τα θέματα δεν ανταποκρίνεται όμως απόλυτα στη σημερινή εποχή παρόλες τις ε, προσπάθειες του παρατηρητηρίου που είναι ιδιαίτερα επενέσιμες βέβαια γιατί η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ασχολείται με αυτά τα θέματα και η Γενική Διεύθυνση Προστασίας των Καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν και συγκεκριμένες ευθύνες, δηλαδή πρόληψη, και πάλι επανένταξη στην κοινωνία για τους χρήστες. Καμιά φορά όμως δεν είναι δυνατόν πρέπει να πούμε να δοθούν κάποια, ε, να δοθεί υποστήριξη στα, στις οικογένειες και η αγορά από ό,τι φαίνεται είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστη. Δηλαδή βλέπουν και χρησιμοποιούν νέα ψυχοτρόπα φάρμακα και νέες δυνατότητες διαρκώς διανοίγονται. Ελπίζω ότι θα υπάρξει σαφής προσανατολισμός ε, για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Θέλω να παρακαλέσω όλους να περιορίζονται σε ένα λεπτό, γιατί διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Όσον αφορά την στοχοθέτηση της προσφοράς από τις αστυνομικές δυνάμεις, ε, τότε βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μπορούν να αυξάνονται οι τιμές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τους μικροχρήστες ε, αντιμετωπίζει, στοχοθετεί η αστυνομία και στην ε, πώληση της ε, λιανικής. Κατά τα άλλα αγνοούν τους ε, εμπόρους που δρούν σε πιο πλούσιες ε, περιοχές και ε, εμπορεύονται ναρκωτικά. Γιατί? Διότι αυτές οι περιοχές είναι εκτός πρόσβασης για την αστυνομία επειδή είναι των ανώτερων τάξεων. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ομιλητές και μετά κλείνει ο κατάλογος. Η κυρία Κέλλερ και μετά ο κύριος Μούλερ και θα τελειώσουμε. Ίσως ε, το έχασα αυτό, θα ήθελα να επεξηγηθεί. Γιατί δεν αναφέρετε το θέμα των ενοπνευματοδών στην έκθεσή σας ή στην ε, γραπτή αυτή διατύπωση. Ίσως ε, ευθύνεστε εσείς, δεν το γνωρίζω αυτό. Ευχαριστώ που είσαστε σύντομοι. Ο κύριος Μούλτερ και μετά Αντζελίλη. Η ερώτησή μου είναι απλή, είναι η εξής. Υπάρχει κάποια σαφής άποψη στο θεσμικό όργανο, στα θεσμικά όργανα για την αποεγκληματικοποίηση της χρήσης ήπιων ναρκωτικών όπως για παράδειγμα η χρήση του ινοπνεύματος των ινοπνευματοδών και αυτή δεν είναι εγκληματική πράξη. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Αντζελίνη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είχα την ευκαιρία την έκθεση μόλις τώρα να την πάρω. Την πήρα μόλις τώρα και έχω μια ερώτηση λοιπόν προς εμάς. Εδώ αναφέρονται smart drugs, σωστό, ευφυή ναρκωτικά, ναι, νέα ναρκωτικά. Θα ήθελα να ρωτήσω, ασχολείται με αυτό το θέμα το smart drugs στο παρατηρητήριο. Είναι από ό,τι φαίνεται μια σοβαρή εμφάνιση, ένα σοβαρό γεγονός αυτά τα smart drugs. Μπορείτε εσείς να τα καλύψετε και σε ποιο πλαίσιο. Και πραγματικά ευχαριστώ και η τελευταία παρέμβαση, ο κύριος Κλοντ Μωράης, όχι, ο, ο επόμενος Μία ερώτηση όχι ε, για ε, τα smart, smart shops και εδώ για το πώς μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, να ετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν τον προβληματισμό των smart shops. Τι γίνεται με τα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτό το φαινόμενο. Δεύτερη ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για το μέγεθος των οικονομιών αυτών. Σας ευχαριστώ λέει ο κύριος Σταβάρες. Κύριε Βίρτσο, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέψετε θα τα πάρω με την σειρά όπως αναφέρθηκαν. Ε, το θέμα για την, το μέγεθος της ε, αγοράς κανάβεως ε, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι δύσκολο Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι 74 εκατομμύρια έχουν κάνει χρήση κανάβεως και υπάρχουν και άλλοι που τα χρησιμοποιούν πιο τακτικά. Έχουμε και ε, κάποια στοιχεία για τους χρήστες. Δεν ξέρουμε όμως ακριβώς το εύρος. Ε, η διακύμαση τιμών διαφέρει από χώρα σε χώρα και η προσφορά, όσον αφορά την προσφορά, χίλιοι τόνοι κατάσχονται κανάβεως ετήσια. Αλλά όπως είπα υπάρχει όλο και πιο γηγενής παραγωγή στην Ευρώπη. Σε σχέση με, αυτό, με αυτούς τους χίλιους τόνους, αν πάρουμε σε ένα χρόνο, τρεις τόνοι τη μέρα βγαίνουν. Έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι ίσως 10% είναι αυτό το οποίο κατάσχεται και θεωρούμε και δεν είμαστε μόνο εμείς αλλά και η Europol και οι αστυνομικέ δυνάμεις θεωρούμε ότι είναι πολύ ευρύτερο αυτό το πλαίσιο αλλά δεν έχουμε ακριβώς ε, τα στοιχεία. Smart shops και legal highs και όλα αυτά τα σύναφη. Αυτό είναι ένας θολός τομέας που δεν θα έπρεπε να βλέπει κανείς ε, μόνο τα νόμιμα ή μη απαγορευμένα ακόμα ε, τέτοιου είδους ψυχότροπα αλλά πρέπει να δει κανείς και την ε, κατάχρηση συνταγών και την δυνατότητα που προσφέρεται ε, στους χρήστες και Θέλω να πω σε σχέση με κάθε χρόνο την ανείχνευση αυτής της, ε, αυτού του φαινομένου των ψυχοτρόπων με τα εθνικά κομβικά σημεία και της ε, Europol έχουμε ε, ε, ας το πω έτσι επικεντρώσει την προσοχή μας σε αυτά και είναι κάτι όπου είναι διαφορετική προσέγγιση από χώρα σε χώρα. Μόλις προανέφερα ότι υπάρχει μία από τις ουσίες η μεθοδρόνη που θα απογορευτεί από το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες ε, μάλλον. Ήδη είναι υπό έλεγχο στις 17 χώρες. Η επιστημονική μας επιτροπή έχει συνεργαστεί. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δράση. Είναι πολύ δύσκολο να δει πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Ενώ σε κάποιες χώρες ε, ε, υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο μέσα στην νομοθεσία κατά των ναρκωτικών, αλλού μέσα στη φαρμακευτική νομοθεσία τα smart shops δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι υπήρξε μια μεγάλη δράση στην Πολωνία τις τελευταίες εβδομάδες όπου μέσα σε μια εβδομάδα έκλεισαν 1100 τέτοια μαγαζιά ε, smart shops όπου μπορεί κανείς να αγοράσει τέτοιου είδους ε, ε, ψυχότροπα φάρμακα και Μπορεί κανείς να, να δει ότι σε σχέση με ένα ε, generic law στην ε, Πολωνία για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ αλλού είναι θέμα αστυνομικών δυνάμεων ε, με παράπλευρες νομικές διατάξεις καταστολής η αντιμετώπιση. Δεν ξέρουμε αν θα στεφτεί με επιτυχία αυτό το μέτρο, αλλά σε κάποιες χώρες αυτά τα smart shops ή όπως και αλλιώς να τα αποκαλούμε, έχουν ε, ε, τέτοιες δυνατότητες ε, στην Πορτογαλία πρόσφατα για παράδειγμα και στα μαγαζιά αυτά πάνε και αγοράζουν κάτι οι πολίτες είναι πολύ εύκολο δίνονται συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα εκεί σε αυτά τα μαγαζιά υπάρχουν οι δυνατότητες αγοράς να αγοράσουν ουσιών που δεν είναι ακόμα απαγορευμένες και επιτρέπεται να τις εμπορεύονται παρακολουθούμε αυτό το θέμα όχι μόνο για να παρακολουθήσουμε τις ουσίες και τα μέτρα και την ανάλυση των μέτρων και των βέλτιστων πρακτικών, αλλά για να αναλύσουμε όλες τις πτυχές και τις νομικές προσεγγίσεις. Αλλά ξεκινάμε νομίζω να βρούμε μια κοινή νομική προσέγγιση για την πρόσβαση αντιμετώπισης αυτού του ε, φαινομένου. Δεν έχουμε από ε, επ' αυτών των θεμάτων που ρωτήσατε κάποια συγκεκριμένη άποψη. Δεν είναι δουλειά μας να έχουμε μια τέτοια άποψη. Αυτό που κάνουμε όμως από την άλλη πλευρά είναι η ανάλυση της κατάστασης, η σύγκριση της κατάστασης ε, στα κράτη-μέλη προσπαθώντας να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ συχνά ξεκινάμε με την απελευθέρωση μια τέτοια τάση. Δεν υπάρχει καμιά χώρα στην Ευρώπη, καμιά κυβέρνηση σε σχέση με την απελευθέρωση των ε, παράνομων ε, ε, τέτοιων ψυχότροπων ουσιών. Είναι διαφορετική η προσέγγιση από χώρα σε χώρα όσον αφορά μικρή ποσότητα για προσωπική χρήση για παράδειγμα που μπορεί να είναι ένα φαινόμενο ανεκτό χωρίς να διώκεται. Αλλά και πάλι υπάρχουν διαφορές πρέπει να πω στον προσανατολισμό ανθρώπων που εξαρτώνται από τέτοιες ουσίες ε, δίνοντας τους ε, συμβουλές για παράδειγμα άλλες ε, φορές προσάγονται στο, στα αστυνομικά τμήματα δεν έχουμε κάποια άποψη επί του θέματος αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς που να έχει φυλακιστεί ή να φυλακίζεται επειδή είναι απλά και μόνο χρήστης ουσιών. Άλλο πράγμα το τι συμβαίνει με τους εμπόρους ναρκωτικών που διώκονται και φυλακίζονται. Με ένα τέτοιο άνοιγμα, α το πω έτσι, μπορούμε να δούμε το τι συμβαίνει με τις ψυχότροπε ουσίες και να δούμε και συγκρίσιμε καταστάσει ε, όπως για την κατάχρηση ναρκωτικών. Αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό το πράγμα πολύ συχνά το ενόπνευμα βρίσκεται στο ε, επίκεντρο ε, προσοχής όσον αφορά την κατάχρηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρτς που είσαστε εδώ ανάμεσά μας και λυπούμε που χρειάστηκε τόσο πιεστικά να τεθούν ερωτήσεις. Οι απομένουσες ερωτήσεις θα πρότεινα να ε, μέσω της γραμματείας να διαβιβαστούν και να υπάρχει δυνατότητα γραπτός να απαντηθούν και στη συνέχεια κύριο Σαχάστεγξα από την εποπτεία των επόπτη προστασίας προσωπικών δεδομένων για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νερφέλτ. Σας ευχαριστώ πολύ που δείξατε και τέτοια ευελιξία και αλλάξατε την ώρα της παρουσίασης. Κατάλαβα ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, οπότε θα είμαι σύντομος. Ο φίλος, ο κύριος Κέτς, παρουσίασε την ετήσια έκθεση 2010. Εμείς ακόμα στην ετήσια έκθεση 2009 είμαστε. Σήμερα το πρωί παρουσιάσαμε τις πρώτες αντιδράσεις μας όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Προστασία Δεδομένων και σίγουρα θα επανέλθουμε. Επί τη ευκαιρία αυτή παρουσιάσαμε και την ετήσια έκθεση. Επί τη ευκαιρία αυτή επίσης θέλω να σας μιλήσω και για τα δύο εδώ. Ας ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Επιτροπής. Το μήνυμα κλειδί σήμερα ήταν ότι η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων είναι πολύ καλό, πολύ σωστό που έρχεται αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να φροντίσει να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία δεδομένων για την περίοδο 2015 και μετά. Και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φανεί φιλόδοξη στις προτάσεις της, προτάσεις που θα υποβάλει στα μέσα της επόμενης χρονιάς. Συγχρόνως όμως, μια που δεν είμαστε στο 2015 ούτε βέβαια και μετά από το 2015, Ας δούμε τι γίνεται τώρα και πώς ε, εφαρμόζουμε τους ε, κανόνες που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας και τι κάνει ο επόπτης προστασίας δεδομένων όσον αφορά τον ε, έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων αυτών και τι κάνουμε όσον αφορά την συνεργασία μας με αυτούς οι οποίοι πρέπει να θέτουν σε εφαρμογή τους κανόνες. Έχουμε καλές εξελίξεις. Οι κύριες τάσεις στον τομέα αυτό και ο Τζοβάνι Μπουταρέλη θα δώσει και περισσότερα παραδείγματα εφόσον έχουμε χρόνο επιθερούμε την κατάσταση όσον αφορά την σωστή εφαρμογή και κάνουμε ελέγχους για τη σωστή εφαρμογή και θα εκδώσουμε και κάτι σχετικά με αυτό. Στον τομέα της διαβούλευσης τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις που ζητούν να διευρυνθεί κάπως το πεδίο εφαρμογής. Υπάρχει πάντως πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους από τα διάφορα κράτη-μέλη. Ο Τζοβάνι θα μιλήσει και για τις προτεραιότητες της επόμενης χρονιάς. Εγώ όμως θέλω να επανέλθω στο πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η δουλειά. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η προστασία δεδομένων είναι κάτι που αποκτώλει και μεγαλύτερη σημασία τελευταία. Είναι κάτι που αναγνωρίζεται σαν σημαντικό και στην Ευρώπη, αλλά και αλλού. Παρόλο που είχαμε την εντύπωση ότι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ, όχι, παίρνουμε θετικά μηνύματα και από εκεί. Και είναι σημαντικό διότι πρέπει να επενδύσουμε σε μια ισχυρή και αποτελεσματική προστασία δεδομένων μέσα σε μια κοινωνία η οποία εξαρτάται όλο και περισσότερο από την πληροφορική. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί και φιλόδοξοι για να ε, διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες τίθενται σε εφαρμογή αποτελεσματικά εντοπίζουμε όλοι τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες δυσκολίες. Η μεγάλη πρόκληση όμως είναι το επόμενο στάδιο. Οι προτάσεις που θα κάνουμε για ένα νομικό πλαίσιο που να καλύπτουν όλο το θέμα και να φροντίζουν να είμαστε αποτελεσματικοί. Τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και το Συμβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι προετοιμάζεστε γι' αυτό και θα μας δοθεί ευκαιρία να προετοιμαστούμε και μαζί. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εκείνη θα κάνει το επόμενο βήμα, που θα αποτελέσει και τη βάση για τη συζήτηση. Το είπα και σήμερα το πρωί, αλλά το επαναλαμβάνω και εδώ τώρα. Εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είσαστε αυτοί που έχουν τον κύριο ρόλο. Οι προκλήσει είναι τεράστιε. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ασφάλματα. Γι' αυτό και οι προτινόμενε λύσει πρέπει να είναι και φιλόδοξε αλλά και αποτελεσματικέ. Δεν έχει νόημα να κοιτάμε πίσω Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά και να επενδύσουμε στην αποτελεσματικότητα. Και αυτό σε πολλούς και διάφορους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη αναρμόνιση στην εσωτερική αγορά και να καθίσουμε ίσως να ξανασκεφτούμε την αρχιτεκτονική του τρέχοντος πλαισίου. Χρειάζονται ευρωπαϊκοί κανόνες που να εφαρμόζονται άμεσα, πιο εύκολα. Ίσως αυτή να είναι μια λύση. Εμείς υπογραμμίζουμε την τεχνολογία, υπογραμμίζουμε αρχές όπως είναι ο ιδιωτικό βίος, η λογοδοσία. Επίσης υπογραμμίζουμε ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Η άποψή μου για την ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ότι έτσι κι η συνθήκη δίνει εντολή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για ένα συνολικό πλαίσιο. Εσείς που είσαστε υπεύθυνοι και για τον προπολογισμό και για την εφαρμογή των κανόνων μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Εφαρμογή των κανόνων σημαίνει και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαίνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα επίσης πρέπει να τηρούν τους παρόντες κανόνες. Πρέπει να φροντίσουμε ιδιωτικό βίο να συμπεριλαμβάνεται σαν έννοια μέσα σε κάθε νέα ρύθμιση. Και πρέπει να συνεργαζόμαστε με διάφορε πλευρέ και διάφορου φορεί. Θα δώσω το λόγο στον Τζοβάνι όμω τώρα, μια που πιέζει ο χρόνο, και μετά, εφόσον έχουμε χρόνο, ευχαρίστω να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Πρόεδρε, όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε σωστά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το 2009. Πρέπει να συνεργαστούμε και με τους συναδέλφους μας στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να υπάρχει ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία δεδομένων παντού. Τα αποτελέσματα του 2009 όσον αφορά την εποπτεία επικεντρώνονται σε τρεις τομείς. Είναι η έλεγχη, ο εντοπισμός των παρατυπιών και η συμμόρφωση. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να εξετάζουμε κατά πόσο τόσα κάνει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για την προστασία των δεδομένων. Έχουμε καλύψει το 2009 περισσότερα θέματα από όσα το 2008, είτε πρόκειτο για υποκλοπές, είτε πρόκειτο για προσωπικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν και δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταφέρει να καλύψουν ακόμα καλύτερα από ό,τι κατά το παρελθόν τις προδιαγραφές για την προστασία δεδομένων. Αλλά υπάρχει περιθώριο για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Γι' αυτό και συνεχίζουμε τους ελέγχους μας σε διάφορα όργανα και οργανισμούς. Και ο αριθμός αλλά και η περιπλοκότητα των προσφυγών που έχουμε Τα δύο τρίτα ε, των ε, προσφυγών που λάβαμε δεν ήταν ε, παραδεκτές. Οι υπόλοιπε έχουν να κάνουν με λεπτά και ευαίσθητα θέματα. Παραβίαση του απόρριτου, υπερβολική συλλογή δεδομένων, παράνομη χρήση τους κλπ. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες προστασίας των δεδομένων παραβιάστηκαν σε 8 περιπτώσεις. Ίσως να είσαστε πιο εξοικειωμένοι με τις νομοδοτήσεις που εκδώσαμε για ευαίσθητα θέματα όπως είναι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και στην έκθεσή μας θα βρείτε και σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την ομάδα εργασίας άρθρο 29. Τέλος. Ποιες είναι οι κύριες προτερότητές μας για το μέλλον. Πέντε σημεία. Νομικό πλαίσιο βέβαια. Ψηφιακή ατζέντα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία μελλοντικός ε, ρόλος των εκ των προτέρων ελέγχων. Συμμόρφωση και τέλος θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε γνωμοδοτήσεις και σχόλια όσον αφορά νομοθετικές προτάσεις σε όλους τους τομείς. Τα υπόλοιπα πράγματα θα τα βρείτε έτσι καλλιώς στο κείμενο. Ευχαριστώ. Ε, έχω μία αίτηση για το λόγο, μία σύντομη ερώτηση εγώ η ίδια. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο τότε η κυρία Κλάσου και η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει μία σύσταση. Έχετε μέτρα τα οποία προτείνετε ε, και το, το ευρωπαϊκό, ε, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση θα πρέπει να την εφαρμόσει. Ε, πόσες φορές όμως πρέπει να επιμείνετε για να μπορέσουν όντως να ισχύσουν τα μέτρα αυτά. Μία ακόμη ερώτηση γιατί η προηγουμένη ήταν πολύ σύντομη. Με συγχωρείτε, η κυρία Λάντφορτ σχετικά με την ε, ε, συνεργασία με την Επιτροπή του άρθρου 29. Ήξερα ότι ε, είχε συζητηθεί, είχε δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει στήριξη για το, την Επιτροπή του άρθρου 29, διότι αν θυμάμαι καλά υπήρχε ε, μία διαφορετική αντιμετώπιση για την ε, ομάδα εργασίας την οποία είχαμε αντιμετωπίσει τότε. Ωραία, αυτό ήταν το πρώτο ήμις της δικιάς μου ερώτηση και το δεύτερο είναι ποιοι είναι οι πόροι για την προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορείτε να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις και στη συνέχεια οι ερωτήσεις μπορούν να τεθούν γραπτός όπως και στην προηγούμενη έκθεση. Βέβαια, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την ανακοίνωση αυτή και να συνεργαστούμε με τον εισηγητή σχετικά με το θέμα αυτό. Σχετικά όμως με την πρώτη ερώτηση θεωρώ ότι αναφέρεται στον μηχανισμό για, την για τον προκαταρτικό έλεγχο. Ε, είχαμε 110 ελέγχους πέρυσι, ε, περίπου 600 αρχικές αξιολογήσεις εφέτος και λέμε ότι αν οι συστάσεις αυτές εφαρμοστούν τότε δεν υπάρχει δυνατότητα παραβίασης. Στη συνέχεια οι ελεγκτές μας ε, ενημερώνουν μετά τρεις μήνες από τις εφαρμογή των συστάσεων αυτών, δηλαδή αν έχουν εφαρμοστεί ή όχι και αν χρειαστεί ξαναεπιμένουμε. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις προχωράμε και διαφορετικά ε, γίνονται ε, επιθεωρήσεις ε, επί των θεμάτων αυτών. Όσον αφορά το άρθρο 29 υπάρχει σίουσα κατά κατάσταση και το μέλλον. Εσείς αναφέρεστε στην ισχύουση κατάσταση. Δηλαδή η τωρινή, το τωρινό σύστημα δεν είναι τέλειο. Μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 29 και της Επιτροπής μας πρέπει να βρεθεί μία λύση. Χρειάζεται κάποια στήριξη και γι' αυτό η βοήθεια δημοσιονομικά του Κοινοβουλίου θα είναι χρήσιμη. Όσον αφορά το μέλλον, η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι σαφής, θέλει να ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα σε εργασίες, να τονίσει το ρόλο της, να ε, επενδύσει στην εφαρμογή τη συστάσεως να καταστήσει τη σύσταση δεσμευτική και εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Μέχρι τότε βέβαια η συνέχιση της ε, στηρίξεώς σας για την Προεδρία της Επιτροπής του άρθρου 29 θα είναι χρήσιμη. Ξέρετε ότι αύριο ε, ε, είναι η τελευταία μέρα να διαπραγματευόμαστε τον προϋπολογισμό για το 2011. Ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά. Αλλά Εάν δεν, τότε ε, οι ελάχιστες συνθήκες για να συνεχίσουμε την εργασία μας του χρόνου πρέπει ε, να καλύπτονται. Δηλαδή ε, εσείς ζητάτε να υπάρξει κάποια αύξηση για να μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα νέα στοιχεία και να συνεχίσουμε και τα προηγούμενα. Εάν όμως η αντίδραση του Συμβουλίου δεν είναι θετική θα υπάρξει πρόβλημα και αυτό είναι σαφές για όλους όσους εμπλέκονται οπότε νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Με υπό την αίρεση αυτή λοιπόν είμαστε τώρα σε θέση εφόσον ε, είμαστε 45 μέχρι 50 του χρόνου θα έχουμε άλλα δύο στοιχεία και θα κάνουμε πάρα πολλές ε, ε, επιθεωρήσεις επισήμως. Ωραία. Μου ελέγχθη τώρα ότι οι διερμηνείς πρέπει να φύγουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι άκουσαν τα τελευταία λόγια σας και σας θα μεταφράσουν αυτά τα οποία θα ε, διαμειφθούν στην Επιτροπή Προπολογισμού ε, προς όφελό σας. Οπότε λύεται η συνεδρίαση όσον αφορά τη διερμηνή.